Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Παρακαλώ να έχω λίγο την προσοχή σας. Γιατί είναι πολύ φορτωμένη η σχεδιάζει αυτές τις δύο μέρες. Δεν έχουμε απλά την τακτική συνεδρία τη Επιτροπή μα, αλλά έχουμε και τη συνεδρία των συντονιστών αύριο. Α περάσουμε όμω πρώτα απ' όλα στην έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Πρώτα απ' όλα έχουμε ζητήσει λάβει κάποια αιτήματα για τροποποίηση του σχέδιου μερισιάς διάταξης. Αυτές τις τροποποίησεις πρέπει να τις εγκρίνετε. Πρώτο σημείο. Έχετε, πρέπει να λάβετε υπόψη τις εξής τροποποίησεις. Αναβολή του σημείου 8. το οποίο αφορούσε την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που συντελείται στη Ρουμανία βάσει του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου. Λάβαμε επίσης συμβαστικές τροπολογίες για την έκθεση ΜΑΚΟΒΕΙ για, για τη δέσμευση και δίμευση των προϊόντων του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσθέσουμε το σημείο αυτό, δηλαδή την εξέταση των τροπολογιών για την έκθεση αυτή. Επίσης το σημείο 4 Eurodac θα πρέπει να περάσει μετά το σημείο 9. Και το 7, ναι, ορίστε. Διάστε μέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν άκουσα καλά είπατε για το σημείο 4 Είπατε ότι θα εξεταστεί μετά το 9. Δεν συμφωνώ. Διότι ακριβώς έχω λιμένες υποχρεώσεις και σε ό,τι αφορά τον κανονισμό 539 και την ομοθετική, το ομοθετικό του καθεστώς, θα ήθελα να συζητηθεί ακριβώς τη σειρά την οποία είχαμε συμφωνήσει προηγουμένως. Πρόεδρος, ακούστε κύριε Διαθετεμέρα, η αναβολή το αίτημα το σχετικό αφορά μόνο την παρουσίαση της κατάστασης των διαπραγματεύσεων της έκθεσης Μακοβέ για το Eurodac. Μόνο για αυτό το σημείο, δηλαδή το σημείο το δικό σας παραμένει στην ημερήσια διάταξη και στο σημείο που ήταν, στη σειρά που ήταν. Επιτρέψατε να ολοκληρώσω πρώτα τις προτινόμενες αλλαγές ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, μίλησα για το 7, μίλα για το 7 μάλλον, Μακιντάρια για την προστασία του ευρώ. Έξι ώρα θα πάει. Και ένα άλλο σημείο θα το δούμε σε κάποιο άλλο, το 33-34 ζητήθηκε αναβολή από τον εισηγητή. Στο 40 για την παρουσίαση της έκθεσης παρακολούθησης εφαρμογής συμφωνίας TFTP κτλ και αυτό θα αναβληθεί για αργότερα. Αλλά, επαναλαμβάνω, αυτά είναι αιτήματα των εισηγητών. Αν εσείς έχετε κάτι να πείτε, κυρία Λάρφορντ, για διαδικαστικό, θα μπορούσατε να μας πείτε για πότε θα συζητηθεί το σημείο που αφορά τη Eurodac, πρόεδρος. Επιμένω, μόνο η έκθεση Μακοβέη δηλαδή την κατάσταση να διαπραγματεύσουν Αυτά θα τα συζητήσουμε μετά το 9. Κάποιες ώρες καθυστέρηση θα υπάρξει μόνο. 12 και 20 δηλαδή, αν το συζητήσουμε. Παρακαλώ, Ματιό. Κύριε Πρόεδρε, τι ώρα είπατε για το σημείο Μακοβέη. Μπορούμε μήπως να το εξετάσουμε το απόγευμα. Θα ήταν προτιμότερο. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Παραλαμβάνω ότι πρόκειται μόνο για την παρουσίαση τη κατάσταση των πραγματεύσεων για την έκθεση Μακοβέη. Για τις δημεύσει, λέει η κυρία Ματιέ. Κοιτάξτε, υπάρχουν περισσότερες της μιας εκθέσει Μακοβέη. Τη δίμευση και δέσμευση. Δέσμευση και δίμευση. Όχι. Αντιθέτως, αυτό που είχε ζητηθεί από την κυρία Μακοβέη ήταν να συμπεριλάβουμε αυτό το σημείο για τις δυσμεύσεις και κατασχέσεις και τα λοιπά στην ημερήσια διάταξη αυτή της συνεδρίας. Έχετε τις προτάσεις τροποποίησης και αυτό που λέμε για την έκθεση ΜΑΚΟΒΕ για τις δεσμεύσεις και δημεύσεις πρώτων εγκλήματος είναι να μπει στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Ματιο... Ναι, συμφωνώ, αλλά να το συζητήσουμε το μεσημέρι λέω και όχι τώρα. Ο πρόεδρος. Νομίζω ότι ε, ρητός η κυρία Μακοβέ ήθελε να συζητηθεί το πρωί. Ζήτησε να μπει για, σήμερα το πρωί. Eurodac όμως, δεύτερη έκθεση Μακοβέ για τη Eurodac. Η σχετική πρόταση είναι να συζητηθεί το σημείο αυτό μετά το σημείο παρθμών 9. 12 και 20. Ματιό. Εντάξει για την ε, Eurodac. Εγώ μιλάω για την άλλη έκθεση για τις δεσμεύσεις και δημεύσεις πρώτων εγκλήματος. Να μπει αυτό το θέμα το μεσημέρι. Γίνεται. Πρόεδρος, γίνεται. Μπορούμε να το προσθέσουμε στην απογευματινή συνεδρίαση, αλλά στι 6 και 4. Το συμφωνείτε? Συμφωνώ, λέει κυρία Ματιέ. Πρόεδρο. Και θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί την έκθεση Μακοβέη για τις δεσμεύσεις δημές πρώτων εγκλήματος. Για να έχουμε χρόνο να προετοιμάσουμε τη λίστα ψηφοφοριών. Γι' αυτό λέγαμε να συζητηθεί σήμερα το πρωί το θέμα καλύτερα και όχι τα απόγευμα για να έχουμε χρόνο. Ματιέ. Τότε εντάξει, το μεσημέρι, λίγο νωρίτερα να το βάλουμε. Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε τι δυνατότητε έχουμε. Πρέπει πάντως να λάβουμε μια απόφαση. Πρώτα απ' όλα κατά πόσο θα συμπεριληφθεί ή όχι το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη, γιατί αυτό προς το παρόν είναι πρόταση. Κυρία Βέμπερ, πρόεδρε, χθε Πολλέ φορές σα είπα ότι τα λέω υποπλήρη σύγχυση για την ημερήσια διάταξη αυτών των δύο ημερών. Μάλλον πιο πολύ για τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Έχουμε σημεία τα οποία από το πουθενά προτείνονται, ούτε η Κομισιόν τα ζήτησε ποτέ, ούτε οι συντονιστές, δεν ελήφθη καμία απόφαση από τους συντονιστές. Γι' αυτά και στο σχέδιο μερισιάς διάταξη που είχαμε λάβει την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ένα σημείο που έλεγε ενδεχομένω προς επιβεβαίωση το οποίο αφορούσε συζήτηση τη εκθέσεως Μακοβέη. Και έλεγε ενδεχομένω, θα ίσως επιβεβαιωθεί. Στο μεταξύ, Ρουί Βάρε, ε, Βό, Χολμάγερ και εγώ καταθέσαμε πρόταση να συζητηθούν τροπολογίε. Φαίνεται κάθε πολιτική ομάδα ε, έχει προβλήματα με τον τρόπο με τον οποίο διατυπωμένε τροπολογίες. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Μπορούμε τέλο πάντων να αποφασίσουμε για την ημερήσια Ξέρετε και εμείς έχουμε ανηλυμένε ε, υποχρεώσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι χρόνος εργασίας, πώς είναι αυτό το πρόγραμμα της συνεδρίασής μας έτσι. Πρόεδρος, κυρία Βέπερ, δυστυχώς ε, δεσμεύουμε από τους ε, κανονισμούς ως πρόεδρος και αν ζητηθεί αναβολή από κάποιον ε, βουλευτή της Επιτροπής μας πρέπει να το θέσω υπόψη σας και η Επιτροπή μας πρέπει να αποφασίσει. Κυρία Βέμπερ, λυπούμε κύριε πρόεδρε, αλλά στις άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου την ημερήσια διάταξη την συμφωνούν και οι συντονιστές, άρα ξέρουν όλοι περί πρόκειται. Πρόεδρος. Και εδώ έτσι γίνεται. Το ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε τακτικές συνεδριάσεις των συντονιστών και συζητούμε τα πάντα. Κάθε θέμα πάρα πολύ προσεκτικά το συστάμε. Ξέρετε, ξέρετε ότι είναι η πιο πολύ άσχολη επιτροπή αυτή εδώ. Και συμβαίνει ενίοτε. Κάποιο εισηγητής από κάποια πολιτική ομάδα δικαιούται να το κάνει άλλωστε, να ζητήσει αναβολή ενό σημείου. Βέμπερ. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Επιμένω να μα πείτε ποιο ζήτησε να μπει αυτό το σημείο στην διάταξη. Πρόεδρο, αν έχετε αντίρρηση, μπορούμε να θέσουμε την πρόταση αυτή σε ψηφοφορία για να δούμε αν θα γίνουν δεκτέ ή όχι τροποποίησει αυτέ. Έχουμε μια ημερήσια διάταξη. Υπήρξαν προτάσει τροποποίηση ημερήσια διάταξη. Σα το λέω προ πενθύμηση. Μέρε, μέρε πριν από τη σημερινή συνεδρίαση. Έτσι συμβαίνει, δεν είναι έτσι. Όχι. Πριν από τρεις εβδομάδες σας στείλανε την ημερήσια διάταξη που έχετε εδώ αναχείρες. Αν υπάρχουν λοιπόν αλλαγές, γιατί ήδη είναι γιατί ήδη οι συγητές ζήτησαν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Λοιπόν, να ψηφίσουμε αν δεχόμαστε ή όχι αυτές τις αλλαγές. Εντάξει, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η κυρία Λάντφορτ. Μα μπορείτε να απαντήσετε το ερώτημά μου αν θα κάνουμε συζήτηση των συμβιβαστικών τροπολογιών για την έκθεση Μακοβέη για τη δίμευση περιουσιακών στοιχείων. Μου λέτε ποια Μακοβέη, μα υπάρχουν χιλιάδες Μακοβέη εκθέσεις αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν είμαι σκιώδης κυρία αλλά με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο λέει η κυρία Βέμπερ νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζουν πολιτικές ομάδες για την έκθεση Μακοβέη για τις δημεύσεις. Εσείς λέτε ενδεχομένως εξέταση των τροπολογιών. Μα αυτό ισχύει. Γι' αυτό σας λέω. Κυρία Λάτφορτ, θέλω να σας εξηγήσω. Εάν θέλουμε να προσθέσουμε αυτό το σημείο εξέταση τροπολογιών για την έκθεση Μακοβέ για τη δίμευση, μπορούμε να το κάνουμε το πρωί μόνο αν αναβάλουμε το σημείο υπαριθμών 8 που αφορά την πρόοδο για τη Ρουμανία. Αν αναβάλουμε τη Ρουμανία μπορούμε να έχουμε καιρό να αντιμετωπίσουμε τη δίμευση. Αλλά σε εσάς εναπόκειται να αποφασίσετε. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Λοιπόν, δέχεστε αυτές τις τροποποίησεις στην μέση ή ου. αν πρόκειται για μια αλλαγή της ημερήσιας διάταξης, πρέπει πάντα να αποφασίσει η Επιτροπή. Δέχεστε να αναβάλουμε το σημείο υπαριθμών 8, την έκθεση για τη Ρουμανία, ναι ή ου. Ε, εντάξει. Το δεύτερο θέμα τώρα. Να προσθέσουμε την έκθεση Μακοβέ στις 11 ακριβώς, γιατί έχουμε αποφασίσει να αναβάλουμε το σημείο 8. Συμφωνείτε να εξετάσουμε την έκθεση Μακοβέη για την ε, δίμευση στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικέ ενέργειε. Εντάξει. Ωραία, συμφωνήσαμε. Όλα τα άλλα σημεία θα αναβληθούν. Γιατί έτσι ζήτησαν οι εισηγητέ. Όλα τα άλλα αναβάλλονται. Λοιπόν, προσπαθήσουμε να βάλουμε έκθεση Μακοβέη. Και τώρα έρχομαι στις ανακοινώσεις. Οι διορισμοί των εισηγητών είναι οι εξής. Σαρτζεντίνη, η εισηγήτρια για την πρόταση οδηγίας για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για έκπληση χρημάτων. Περιλαμβάνει και από τρομοκρατικές ενέργειες. Και η κυρία Σαρτζεντίνη είναι εισηγήτρια για το θέμα αυτό. έγκριση των πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσει οι οποίες θα διατυπωθούν, θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Πάμε στο πρώτο ουσιαστικό στοιχείο στην ημερήσια διάταξη που είναι το σημείο υπαριθμών 4. Κατάσταση πραγμάτων για τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Έχουμε καταρχήν την έκθεση δια Μέρα για τις προξενικές θεωρήσεις όταν περνάμε τα εξωτερικά σύνορα. Μετά έκθεση Αντωνέσκου για τις ε, ποινικέ διαδικασίες και την έκθεση Γιγιόμ για τις διαδικασίες στα κρατημέλη για την ε, παραχώρηση ή την απόσυρση διεθνούς προστασίας. Δίνω λοιπόν καταρχήν το λόγο στους συζητητές να παρουσιάσουν την κατάσταση των διαπραγματεύσεων ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρομαι στον κανονισμό, στην τροποποίηση του κανονισμού 539. Και ξεκινώ με τον ίδιο τρόπο <clears throat> με τον οποίο θα τελειώσω. Σου απειτερημόντο, in Ρέ Είναι ισχυρό το περιεχόμενο λοιπόν αυτού του νομοθετήματος. Αυτό είναι το ουσιαστικό θέλω να πω για τη στάση του Συμβουλίου. Όπως έχει εκφραστεί από την Προεδρία του Συμβουλίου, το Συμβούλιο έχει δράσει με έναν τρόπο απαράδεκτο. Τώρα, ακούγεται τώρα. Έχουν ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι απόλυτα απαράδεκτος για το Κοινοβούλιο και δεν δείχνει τον παραμικρό σεβασμό για τις αρμοδιότητες του, του Κοινοβουλίου. Η κατάσταση λοιπόν στην οποία βρίσκεται αυτή η πρόταση σε νομοθετικό επίπεδο είναι η εξής. Μετά από τα τελευταία γεγονότα και μετά από την ανάληψη της Προεδρίας από την Ιρλανδία μέχρι την τελευταία μου παρουσία εδώ που σας έδωσα μία ενημέρωση για την κατάσταση των πραγμάτων και για την εξέλιξη η οποία έχει υπάρξει, καθώς και για τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε μέσα στα πλαίσια της, νομοθε... της διαπραγματευτικής εντολής που μου έχει δώσει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έχουν λάβει χώρα διάφορα γεγονότα που είχαν σαν αποτέλεσμα η συζήτηση για αυτή την έκθεση που προβλεπόταν στην αρχή για τις συνεδριάσεις μας το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο αναγκάστηκε να αποσυρθούν από την ημέρηση διάταξη. Την τελευταία μου παρουσίαση αυτής της έκθεσης Σα υπενθύμισα ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο σε σχέση με το θέμα της αμοιβαιότητα. Που θα έπρεπε να βασιστεί σε χρήση και κατεχώρηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων. Στι 19 Δεκεμβρίου πρόκειται να γίνει αυτό στην Κορεπέρ, η συμφωνία η τελική. Αλλά επειδή ήταν φανερό ότι δεν θα υπήρχε η απαραίτητη ομοφωνία στο Συμβουλίο και επειδή η Κομισιόν αντετίθετο, το ίδιο το Συμβούλιο αποφάσισε να αποσύρει το θέμα αυτό από την ημερήσια διατάξη της Κορεπέρ. Μετά από όλα αυτά, εγώ μαζί με τους όλες συζητητές συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει και εμείς να προβούμε σε περαιτέρω προβληματισμό για τα επόμενα βήματα και να αποσύρουμε το θέμα αυτό από την ημερήσια διάταξη. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο αρνητική ήταν και επικίνδυνη η στάση του Συμβουλίου γιατί επί τη βάση του εγγράφου του Δεκεμβρίου που περιείχε τις συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί με τις προηγούμενες προεδρίες, τελευταία στιγμή ορισμένες χώρες στα πλαίσια του Συμβουλίου έδειξαν δισταγμούς για συγκεκριμένα στοιχεία της πρότασης αυτής. Και αυτό δεν αφορά μόνο το μηχανισμό αμοιβαιότητος, αλλά και το μηχανισμό αναστολής, ο οποίος είχε στο παρελθόν εγκριθεί με ομοφωνία. Όπως είπα, τον Ιούνιο του 2012 η Ποδανική προεδρία είχε γίνει δεκτή η διαδικασία αναστολής. Μετά από την ρήξη αυτής της συμφωνίας, η Ιλλανδική Προεδρία έκανε μια συνεδρίαση των εμπειρογνωμόνων για τα θέματα αυτά το Φεβρουάριο, οι οποίοι συζήτησαν για το μηχανισμό αμοιβαιότητας. Ως αποτέλεσμα παρουσιάστηκε ένα τελείως διαφορετικό κείμενο από τα συμπεφωνημένα και αυτά που είχαν τύχει διαπραγματεύσει στο παρελθόν. Το νέο αυτό κείμενο περιέχει εν συνόψη την αυτόματη επανεισαγωγή, αυτόματη τρόπος του λέγει δηλαδή, γιατί αυτός ο αυτοματισμός που περιέχεται στο νέο κείμενο έχει ένα χρονικό ορίζοντα τεσσάρων ετών, τεσσερ, τεσσάρων και ημίσεως έτους μάλιστα. Η πρόταση αυτή είχε απορριφθεί πλήρως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από ό,τι ξέρουμε και από την Κομισιόν έχει απορριφθεί. Με αυτό το νέο πλαίσιο που δημιουργεί η νέα Προεδρία και που αντανακλά μόνο τη θέση της Προεδρίας και όχι όλου του Συμβουλίου προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις δυνατότητε μιας νέας συμφωνίας στα εξή θέματα. Για τα θέματα της αμοιβαιότητα, να επανέλθουμε στο κείμενο το οποίο είχε συμφωνηθεί το Δεκέμβριο, δηλαδή να υπάρξει μια μεικτή χρήση εκτελεστικών και κατεχώρηση πράξεων και στα θέματα της αναστολής το να διαγραφεί κάθε μνήα ποσοστών και να χρησιμοποιηθεί ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών και όχι 4,5 ετών. Η Προεδρία, η Ιρλανδική Προεδρία θεωρεί λαθασμένα κατά την άποψή μου ότι θα μπορέσει να πάρει την ε, υποστήριξη των κρατών που αντιτίθενται σε αυτό το έγγραφο εάν υπάρξει μια συμφωνία για την αναστολή και για τα θέματα της αμοιβαίωτο. Αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Όλο το έργο το οποίο έχει φέρει σε πέρα στο Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά ήταν ευρύτατο έγινε με και επικοδομητικό τρόπο και γι' αυτό πρέπει να εκφράσω την απόλυτη μας απογοήτευση εναντί αυτής της αλλαγής τάσης του Συμβουλίου που δεν καθιστά την επίτευξη συμφωνίας δυνατή. Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε η νομοθετική αυτή πρόταση πριν από 21 μήνες είχαμε Διαπραγματεύσουμε την Πολωνική, Δανική, Κυπριακή και τώρα ιλλανδική Προεδρία. Κάναμε πολλού τριγωνικού διαλόγου, συναντήσει των σκιωδών εισηγητών, συζητήσει σε τεχνικό επίπεδο, σε επίπεδο συνεργατών, σε επίπεδο νομικών συμβούλων. Πάρα πολλέ συνεδριάσει μαζί με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και με τη γραμματεία τη Επιτροπή ΛΥΜΠΑ. Και επιπλέον <clears throat> μια συνεδρίαση που οργάνωσα και εγώ ίδιο μαζί με την. έκανα ο ίδιο μάλλον με την Επίτροπο Μάλστρομ στην τελευταία Ολομέλεια και συγχρόνω πρέπει να αναφέρω και την επιστολή που αποστήλαμε στην κυρία Μάλστον και στην Προεδρία του Συμβουλίου και στα κράτη-μέλη που είχε υπογραφεί από όλου του σκιώδει εισηγητές. Όλα αυτά που σα είπα καταδεικνύουν πόσο μεγάλη ήταν η δική μας προσπάθεια για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική για όλου συμφωνία. Και επίση ήταν συνεκτική και επικοδομητική η στάση τη Κομισιόν. Δεν είχαμε πάντα την ίδια θέση μαζί με την Κομισιόν για τα ζητήματα αυτά, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Κομισιόν κράτησε μια στάση η οποία ήταν συνεκτική και συνεπής. Βέβαια αυτό μπορεί να συνάδει με διαφορές που έχουμε με την Κομισιόν, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ποια είναι η θέση της Κομισιόν. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το ίδιο και για το Συμβούλιο, του οποίου η θέση ήταν ε, αντιφατική και συνεχώς μεταβαλλόμενη. Αυτά τα οποία αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν με τη Δανική Προεδρία δεν ίσχυαν για την Κυπριακή Προεδρία και αυτά που συμφωνήθηκαν υπό Κυπριακή Προεδρία δεν γίνονται δεκτά υπό Ιρλανδική Προεδρία. Όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, θεωρείται ότι είμαστε ενήλικες, ότι νομοθετούμε για το καλό της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η στάση του Συμβουλίου δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι από τη μία πλευρά το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αμοιβαιότητα και από την άλλη πλευρά παρουσιάζουν προτάσεις τόσο απαράδεκτες όσο αυτές που έχουμε ενώπιον μας αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να σας δώσω σαν παράδειγμα αυτών των αντιφάσεων το εξής. Σημείο 3α, το οποίο είναι δεκτό από το Συμβούλιο, λέει τα εξή. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αντιδράσουν από κοινού δίνοντας μια ενιαία απάντηση στην κατάσταση, σε μια κατάσταση που αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα πρέπει να επιτρέψει οι πολίτες της να μην αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Η πλήρης ε, απελευθέρωση στον τομέα των προξενικών θεωρήσεων είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να πριτανεύει στις σχέσεις της με τρίτες χώρες για να μπορέσει να εδραιώσει και την συνεκτικότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θαυμάσια. Πώς δέχεσαι αυτές τις αιτιολογικές σκέψεις και μετά να έρχεσαι με μια εξαιρετικά ελαφριά προσέγγιση αυτοματισμού που, που στηρίζεται στα 4,5 χρόνια και αν μου επιτρέπετε τη, την ηρωνία σχεδόν όσο κρατάει η θητεία της Επιτροπής όπως σωστά σχολίασε η κυρία Βέμπερ. Συνεχίζει κατόπιν το κείμενο. Η εφαρμογή εφαρμόζεται, αναφέρεται στο Συμβούλιο μετά την με για να εξασφαλιστεί η σωστή εμπλοκή των κρατών μελών στην λειτουργία του μηχανισμού αμοιβαιότητας λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα που έχει η διακοπή της χορήγησης θεωρήσεων και οι οριζόντιες επιπτώσεις της για τα κράτη-μέλη του εταίρου στον χώρο Σέγγεν, προσοχή σε αυτό, και για την Ένωση συνολικά. Ιδίω για τις εξωτερικές τη σχέσεις τελειώνω την παράθεση. Από την αρχή των διαπραγματεύσεων όλοι συμφωνήσαμε ω προ τη σπουδαιότητα και τον λεπτό χαρακτήρα του περιεχομένου τη εκθέσεω. Έχει ιδιαίτερη πολιτική ευαισθησία που επηρεάζει όχι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά και τα λοιπά θεσμικά όργανα, ιδίω δε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε συνομοθέτος και δεν πρόκειται να δεχθούμε να μας αποκλείουν από την νομοθετική δραστηριότητα που μας αναφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Η πρόταση του Συμβουλίου αποκλείει το Κοινοβούλιο ως εάν η αρμοδιότητα αυτή δεν ήταν δική μας. Δεδομένης της καταστάσεως, χθε το βράδυ είχαμε την τελευταία συνάντηση ε, των σκιωδών εισηγητών. Ομόφωνα αποφασίσαμε να προτείνουμε στους συναδέλφους στην Επιτροπή να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια στις 20 Μαρτίου. Ζητήσαμε από τις υπηρεσίε μας να ετοιμαστεί μια νέα συμφωνία συνένεσης που θα αντικατοπτρίζει την πλιστάκης εκπεφρασφής αφέση του Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο της ισότητας και της διοργανικής συνεργασίας. Πρόεδρε, είπα ότι θα τελειώσω όπως ξεκίνησα. Μας λυπεί το ότι το Συμβούλιο παρουσιάζει μια παράνομη πρόταση, όχι υποθετικά παράνομη, παράνομη το λέω, και προσβλητική για το Κοινοβούλιο. Παρακαλώ να είναι σαφές αυτό. Θα επανεξετάσουμε με την ψηφοφορία το θέμα της αναστολής, ούτω ώστε κατά πάσα πιθανότητα να την συνδέσουμε με την υιοθέτηση εξουσιοδότηση πράξεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Διευθυντεμέρα. Πληρέστατη ε, παρουσίαση. Δεν έχουμε χρόνο κατάσταση των διαπραγματεύσεων είναι. Δεν πρέπει να υπάρχουν συζητήσεις. Βλέπω ωστόσο ότι σηκώθηκε το χέρι, το χέρι της κυρίας Τεγιόγκ. Δύο λεπτά αν θέλετε για να μιλήσει το Σκιώδης εισηγήτηρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι. Νομίζω εξακολουθεί να υπάρχει ανοιχτό αυτό το θέμα. Υπήρξε αυτή η προσπάθεια να υπάρξει μια σύμβαστη λύση, αλλά όπως είπε και ο κ. Δίας Δεμέρα, απέτυχε αυτή η προσπάθεια και το κάνει σαφές ο κ. Ε, Δεμέρα. Αυτό είναι μια παράδεκτη στάση του Συμβουλίου και είναι μια στάση αντιφατική με τις προηγούμενες θέσεις του. Είναι φανερό ότι το Συμβουλίο δεν είναι αξιόπιστο εταίρο και δεν έχει την πρόθεση να διαπραγματευτεί μαζί μα σε επίπεδο ειλικρίνειας είναι φανερό ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις για τα αντικείμενα αυτά. Το Κοινοβούλιο έχει κατανοήσει αυτή τη διαδικασία ως μια μορφή αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά τα κράτη-μέλη θέλουν να έχουν αυτοί όλα τα ατού στα χέρια τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε τονίσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η διαδικασία της ομοφωνίας είναι υπερβολικά επαχθής. Αυτό δεν θα πρέπει όμως να την χάνει εκμετάλλευση από τα κράτη-μέλη. Εμείς μετά από όλες αυτές τις ε, αρνητικές αυτές εμπειρίες θα πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ προσεκτικοί στις περαιτέρω συζητήσεις με το Συμβούλιο και με την Ιρλανδική Προεδρία. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ότι θα ξεκινήσουν οι προεκλογικέ εκστατείε σε διάφορε χώρε, ιδίω στη Γερμανία, και δεν θα πρέπει να αφήσουμε να είμαστε αντικείμενο εκβιασμών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για την ανακατονομή των εξουσιών. Πρέπει λοιπόν να, προβλημα... να μας προβληματίσει το θέμα αυτό. Αν τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να προχωρήσουμε σε μία συμφωνία, θα πρέπει και εμείς να σταματήσουμε να υποστηρίσουμε τις συμβαστικές λύσεις που έχουν ε, ευρεθεί στο παρελθόν και θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα από την αρχή. Κυρία Βέμπερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι σπάνιο στο Κοινοβούλιο όταν υπάρχει συνένεση για κάτι, αλλά για αυτή την έκθεση σίγουρα υπάρχει συνένεση και αυτό εν πολλής χάρη και στην πολύ καλή δουλειά του εισηγητού μας, κ. Ντίας Ντεμέρα. Χτες συμφωνήσαμε να ακολουθήσουμε πλήρως την γραμμή που προτείνει. Είναι απαράδεκτο το Συμβούλιο να μπορεί να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο και να μην υπάρχει αντίδραση από πλευράς μας όπως αρμόζει. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντίας Ντεμέρα για την στάση του και τον υποστηρίζω. Και η ομάδα μας δεν ήταν ευτυχής με την συμβιβαστική πρόταση για το μηχανισμό αναστολής. Εξού και η αποχή μας στην ε, ψηφοφορία προσανατολισμού. Βλέπετε ότι δεν λειτουργήσε τώρα αυτός ο συμβασμός και πρέπει να επανέλθουμε ενισχύοντας την θέση μας επανεξετάζοντας τις, ε, το ενδεχόμενο σύνδεσης κατεξιδωτών συμπράσεων με αναστολή. Υποστηρίζω την έκθεσή μας λοιπόν και το είπα και χθες στους ε, σκιώδεις. Κύριε Ένστ. Χθες κάναμε σαφές τις συνεδρίες που κάναμε ποια θα ήταν η θέση μας για τα θέματα αυτά πρέπει να πω ότι εγώ προσωπικά ότι εγώ υποστηρίζω απόλυτα τον εισηγητή για τα θέματα αυτά και υποστηρίζω και την θέση την οποία παρουσίασε, είναι ένα τεράστιο, ένα ουρανο, ουρανόμικες σκάνδαλο το γεγονός ότι το Συμβούλιο μας αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό πια μεγαλύνει. Είναι πέντε χρόνια που το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο, οι εξουσίες της Κομισιόν περικόπτονται και ουσιαστικά αποκλείει τη δυνατότητα της να επηρεάσει αυτή την πρόταση. Καταλήγουμε λοιπόν σε καταστάσεις που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πια και απλώς θα πρέπει να το καταγράψουμε αυτό το γεγονός και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα πρέπει να δράσουμε όταν συγκρουόμαστε με πλάκες γρανίτη από την πλευρά του Συμβουλίου συνέχεια. Όλοι οι κανονισμοί του Σέγγεν οι οποίοι, οι οποίοι βρίσκονται σε συζήτηση αυτή τη στιγμή μας βλέπουν να προσκρούμε πάλι σε αμετακίνητα τείχη από την πλευρά του Συμβουλίου. Στις 20 Μαρτίου θα γίνει η ψηφοφορία για τα θέματα αυτά, αλλά εγώ δεν βλέπω καμία άλλη δυνατότητα από τη δική μας πλευρά, γιατί πραγματικά 1,5 χρόνο διαπραγματευόμαστε και όλα αυτά τα που έχουμε διαπραγματευτούν έχουν σβηστεί τώρα με μια μονοκονδυλιά. Εγώ δεν μπορώ να πιστεύω και να ελπίζω ότι θα υπάρξει κάτι το οποίο θα αλλάξει με τι 20 Μαρτίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε λοιπόν αυτή την κατάσταση και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, ευχαριστούμε του κοιόδη εισηγητέ και τον εισηγητή. Έκαναν πολύ σαφεί δηλώσει. Οριστική, τελεσίδικη είναι νομίζω η θέση του Κοινοβουλίου με σπάνιο επίπεδο συμφωνίας για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Έχουμε το ακόλουθο σημείο τώρα. Παρακαλώ, σύντομα. Γιατί δεν πρέπει από το πρωί να καθυστερούμε. Ο κύριος Αντωνέσκου για την πρόσβαση δικηγόρων σε ποινική... Η κυρία Αντωνέσκου για την πρόσβαση δικηγόρων σε ποινικέ διαδικασίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ξεκινώ θυμίζοντας τους συναδέλφους ότι το σχέδιο οδηγίας θέτει ελάχιστους κανόνες για τα δικαιώματα των υπόπτων σε ποινικέ διαδικασίες ανά την Ένωση, δίνοντάς τους το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο και επικοινωνία με τρίτα μέρη όπως ε, προξενικές αρχές, τον εργοδότη τους, συγγενή το ψηφίσαμε τον Ιούλιο. Το Συμβούλιο έχει μια γενική, λάβει μια γενική προσέγγιση, έλαβε μια γενική προσέγγιση στις, ε, τον Ιούλιο του 12. Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο ξεκίνησαν τον ε, Σεπτέμβριο. Είχαμε τρεις τριλόγους υπό την Κυπριακή Προεδρία και μια σειρά συναντήσεων με, τεχνη, με συζητητές και τεχνικές συναντήσεις. Δεν μπορέσαμε να ε, πετύχουμε συμφωνία με την Κυπριακή Προεδρία. Ξεκινήσαμε με την Ιρλανδική Προεδρία τον Ιανουάριο με δύο τριλόγους μέχρι τώρα. Το τελευταίο έγινε χτες. Υπήρξε μια σειρά συναντήσεων με τους σκιώδεις συζητητέ και μια σειρά επίση τεχνικών συναντήσεων. Πρέπει να σας πω ότι συζητώνται όλα τα άρθρα τη οδη... όλα Είναι έντονη συζήτηση, επικοδομητική θα έλεγα, επήλθε πρόοδο, σημαντική πρόοδο. Μην ξεχνάτε ότι η αρχική θέση του Κοινοβουλίου ε, διέφερε από την αρχική θέση του Συμβουλίου. Νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό επί μια σειρά θεμάτων. Ταυτόχρονα ωστόσο υπάρχουν διστάμενες απόψεις για συγκεκριμένα σημεία. Ευχαριστώ τους σκιώδη εισηγητές, διότι όλοι δούλεψαν ε, εξ αρχής με την έκθεση και το προσωπικό μας βοήθησε. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι τεράστια και είναι πολύ ευαίσθητα. Η σπουδαιότητα της έκθεσης επίσης είναι καθοριστική και θα ήθελα να σας πω ότι Δουλέψαμε πολύ καλά στο Κοινοβούλιο και ελπίζω στο μέλλον να επέλθει συμφωνία με το Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή ούτως έχουν τα πράγματα, δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί λέτε ότι δεν έχουμε χρόνο. Οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες των ε, προβλημάτων που υπάρχουν ανά άρθρο. Είμαι έτοιμη ωστόσο να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση μου ζητηθεί. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος ο γιατί που θέλει το λόγο. Όχι. Κύριε Λάτφορντ. Εξαιρετική δουλειά κάνει κύριε Αντωνέσκο, αυτό μόνο θέλω να πω. Μας βάζει όλους στη συζήτηση και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τις διαπραγματεύσεις και με εξαιρετική υποστήριξη από την Γραμματεία. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Και ήσασταν και σύντομοι. Κύριε Γκυγιόμ, για την έκθεσή της για τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας. Θα είμαι σύντομη και εγώ κύριε Πρόεδρε, στο βαθμό του δυνατού. Θέλω να σας αναφέρω ότι για την έκθεση αυτή έχουμε κάνει τρεις τριγωνικούς διαλόγους. Ο τελευταίος ήταν στις 17 Δεκεμβρίου όπως ε, ήθιστε τίποτα δεν ισχύει αν δεν έχουν συμφωνηθεί όλα τα θέματα αλλά η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα περισσότερα θέματα βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στη συμφωνία την στρατηγική εξισορρόπησης και σε επίπεδο διαδικασιών σεβασμού των δικαιωμάτων και διατήρησης της διαδικασίας λήψης απόφασης και συγχρόνως την παρακολούθηση των πολιτικών, δηλαδή να έχουμε μια πολιτική που καλύπτει και τα δικαιώματα των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και πάντα μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πνεύματος. Παραμένουν εκρεμή δύο σημεία διαπραγμάτευσης, τα οποία λιγάκι μπεπλεγμένα για δύο άρθρα το άρθρο 24 για τα θύματα βασανιστήριων και το 25 για τους μη συνοδευόμενους ανήλικους. Επίσης, κάτι το οποίο είναι επίσης επίμαχο, είναι η ιδιαίτερη μεταχείριση που θα πρέπει να επιφυλάξουμε σε αυτές τις δύο κατηγορίες ευαλώτων ατόμων μεταξύ αυτών που ζητούν τη διεθνή προστασία. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται ενώπιόν μας, εν συνόψη, είναι κατά πόσο ναι ή όχι αυτές οι ιδιαίτερες ομάδες μπορούν να απολαμβάνουν μια μεταχείριση η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους σε διαδικαστικό επίπεδο και περιμένουμε την απάντηση του Συμβουλίου σχετικά. Μετά από τον τελευταίο τρίλογο, το Κοινοβούλιο παρουσίασε προς το Συμβούλιο μια νέα πρόταση διατύπωσης για τα άρθρα αυτά, 24 και 25, η Ιρλανδική Προεδρία, την οποία χαιρετίζω εδώ και η οποία έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό με μεγάλη σοβαρότητα προσπαθεί μαζί με τις εθνικές αντιπροσωπείες να καθορίσει τη θέση του Συμβουλίου για τα δύο αυτά θέματα και περιμένουμε τις αντιπροτάσεις που θα διατυπώσει το Συμβούλιο. Ελπίζουμε ότι θα βρίσκονται στο ύψος των προσδοκιών μας και επομένως τα κείμενα αυτά θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε μια αποτελεσματική απόφαση και θα διατηρήσουν την ποιότητα που πρέπει να έχουν αυτά τα νομοθετήματα. Και πάλι πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο να δικαιολογήσουμε μια προσέγγιση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις απαραίτητες απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε στα προβλήματα αυτών των δύο κατηγοριών ευαλώτων ατόμων, πιο ευαλώτων από όλα τα ευάλωτα άτομα. Περιμένουμε φυσικά τις προτάσεις του Συμβουλίου που θα τις εξετάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον μαζί με τους σκιώδεις συζήτητες και ελπίζω θα μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατό να οργανώσουμε ένα τριγωνικό διάλογο ακόμα για να περατωθούν οι διαπραγματεύσεις για το κείμενο αυτό το οποίο ξέρετε ότι είναι ήδη πολύ πολύπλοκο. Ευχαριστώ κυρία Γιγιόμ. Η κυρία Βίξτρομ από τους σκιώδεις συγητές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τη Σιλβή που νυχθημερών έχει εργαστεί για αυτό το τόσο πολύπλοκο θέμα και βλέπουμε τελικά φως στο τέλος του τούνελ και μπορώ να υποστηρίξω απόλυτα το έργο που κάνετε ως εισηγήτρια ιδίως για τα θύματα βασανιστήριων και τους ασυνόδευτους ανήλικους. Μιλάμε για τα άρθρα 24 και 25. Για τις δύο αυτές ευάλωτες ομάδες πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι αυτές οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή τα πιο ευάλωτα άτομα στο ευρωπαϊκό έδαφος σήμερα. Πρέπει να τύχουν λοιπόν προστασία και γι' αυτό υποστηρίζω όλη την προσπάθεια που έχετε καταβάλει για το θέμα αυτό και θα ήθελα να σας παροτρύνω να παροτρύνω μάλλον την Προεδρία του Συμβουλίου και το Συμβούλιο να πάρει όλα αυτά τα θέματα στα σοβαρά και να κατανοήσει την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Γιατί για το θέμα αυτό είμαστε ενωμένοι και υποστηρίζουμε ε, διαρρήνει τη θέση της εισηγήτριας. Για το συνολικό πακέτο τώρα. Κοντεύουμε να φτάσουμε μια συνολική λύση. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε υποσχεθεί στους Ευρωπαίους πολίτες ήδη από το 1999. Είναι καιρός λοιπόν να καταλήξουμε σε μία λύση. Το ταχύτερο λοιπόν που θα κλείσει αυτό το θέμα, το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο, μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, έχοντας ακούσει τις παρουσιάσεις αυτές για τα θέματα αυτά, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5 που είναι η πρώτη έκθεση για την αγορά ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την παρουσίαση του κυρίου Wolfgang Goetz. ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Ναρκομανία, που συνεργάζεται με την Ευρωπόλ και έχουν προβεί σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς ναρκωτικών, της διανομής ναρκωτικών, της τοξικομανίας με διάφορες προτάσεις τις οποίες θα μας υποβάλουν. Και μετά την παρουσίαση θα έχουμε χρόνο για ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων για τα επόμενα 45 λεπτά. Ο κύριος Γκέτς λοιπόν έχει το λόγο. Καταρχήν και μετά ο κύριος Ερτινγκ ο οποίος είναι ο αναπληρωτής διευθυντής για τα θέματα σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Δίνω καταρχήν το λόγο στον κύριο Γκέτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα σήμερα μαζί με τον συνάδελφό μου την Europol να σας παρουσιάσουμε τα πορίσματα της πρώτης έκθεσης ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την αγορά ναρκωτικών, κάτι που μας είχε αναθέσει πριν από κάποιες ε, εβδομάδες η Επίτροπος Μάλστρομ. Europol και ε, εμείς εδώ και 10 χρόνια εργαζόμαστε για το ζήτημα αυτό. Πολλές είναι οι δημοσιεύσεις που έχουν ήδη δει το φως. Και σήμερα θέλουμε να προβούμε σε μια στρατηγική ανάλυση της αγοράς ναρκωτικών συνολικά. Και βέβαια η συνεργασία των δύο οργανισμών είναι ακριβώς αυτή που εξασφαλίζει ε, μια απάντηση ε, η οποία μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία δεκαετία ο κόσμος έχει βιώσει μια περίοδο ε, έντονων αλλαγών λόγω της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής πρόοδου αλλά και του τρόπου με τον οποίο ε, οι άνθρωποι εργάζονται, συναναστρέφονται ένας στον άλλον. Ε, έχουν αλλάξει τρόποι αυτοί και αυτό επηρεάζει και την αγορά των ναρκωτικών σήμερα. Αντιμετωπίζουμε μια τελείως διαφορετική ε, κατάσταση στον χώρο, στην αγορά αυτή και πρέπει να τα ανταποκριθούμε και εμείς στις νέες πραγματικότητες. Το θετικό είναι ότι ο συνδυασμός δράσεων αυστηρών και στον τομέα της προσφάσεως και στον τομέα της ζήτησης οδήγησε σε μείωση προβλημάτων σχετιζόμενο με την ηρωίνη στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα καλό επιχείρημα σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν επηρεάζουν θετικά οι προτάσεις και οι πολιτικές για την καταπλήρωση σκοτικών. Όμως, ό,τι αφορά τις συνθετικές ουσίες και την κοκαίνη, ε, βλέπουμε να προσλαμβάνουν μεγαλύτερη, πιο υψηλή θέση στην αγορά ε, και βλέπουμε τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν πολλές, περισσότερες της μιας ουσίες ή υποκατάστατα ε, ουσιών για να αντιμετωπίσουν τη θεσιμότητα, τη τιμή ή την υποτιθέμενη, ε, ε, όπως να αντιλαμβάνονται, ποιότητα. Δεν μπορούμε πλέον όμως ε, να βλέπουμε μεμονωμένα τα ναρκωτικά, αλλά να υιοθετήσουμε μια πιο συνολική προσέγγιση σε, Ευρωπαϊκή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα το δείτε και στην έκθεσή μας. Είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε αυτή τη νέα προσέγγιση και σε ό,τι αφορά και τα νόμιμα λεγόμενα ναρκωτικά, τα οποία ε, πλέον μπαίνουν στην αγορά με υποτιδευμένους τρόπους ε, και πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. 73 νέες ουσίες κοινοποιήθηκαν στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που ε, λειτουργούμε από κοινού εντός του 2012, από 49 του 2011 220 δε ουσίες από το 2005 και μετά έχουν κοινοποιηθεί σε αυτό το σύστημα. Μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα ε, είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτά τα νόμενα ναρκωτικά, προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν χημικά κοκτέιλ, ε, μάλλον περίπλοκα κοκτέιλ με πολλά χημικέ ουσίες. Αυτά βγαίνουν και στο εμπόριο με ελκυστικές συσκευασίε, ε, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι νέοι να δοκιμάζουν τις ουσίες αυτές, για τις οποίες ξέρουν πάρα πολύ λίγα πράγματα. Το διαδίκτυο είναι ένα όχημα καινοτομία στο τομέα αυτό και είναι και ένας νέος εικονικός τόπος ε, αγοράς, αν θέλετε. Άρα είναι παγκοσμιοποιημένο το πρόβλημα. Η διάδοση ναρκωτικών γίνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι παλιά. Τα τελευταία χρόνια στο έκπλην του έχουμε ε, εντοπίσει 700 νέα ε, στόπους πώλησης διαδικτυακούς Πολλούνται λοιπόν από το διαδίκτυο τα ναρκωτικά αυτά σε πελάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθω στην κάναβη. Η κάναβη δείχνει ε, πολύ καλά ε, τις εξελίξεις σήμερα στην αγορά των ναρκωτικών. Όπως και με τα συνθετικά ναρκωτικά βλέπουμε ότι παράγεται πλέον το ναρκωτικό κοντά στους ε, καταναλωτές, κοντά στους πελάτες τους. Και αυτό είναι μια τάση που θα γενικευθεί και στο μέλλον. Σήμερα η κάναβη παράγεται σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη και συχνά καλλιεργείται εντατικά ε, με υψηλή τεχνολογία. Θα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι η κάναβη που παράγεται με τις μεθόδους αυτές ε, έχει μεγάλη ε, δύναμη, ισχύ και ενδεχομένως είναι και πολύ πιο επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία. Η παραγωγή της κάναβης σχετίζεται με την ζήτηση στην Ευρώπη. 2.500 τόνοι κανάβες καταναλώνονται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. 18 με 30 δις είναι η αξία. Με βάση τις εκτιμήσεις, η μεγαλύτερη αγορά για την κάναβη είναι στην Ιταλία, την Ισπανία και την Γαλλία. Και επίσης και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. για την κάναβη που καπνίζεται σε μορφή χόρτου βλέπουμε να αυξάνεται η κατανάλωση και η παραγωγή και όλα αυτά μας ε, δημιουργούν πρόβλημα. Η κοκαίνη είναι η δεύτερη πιο συχνά ε, παραγόμενη. Η Ισπανία, Πρωτογαλία είναι τα σημεία εισόδου κυρίως για την κοκαίνη στην Ευρώπη. Νοτιοδυτική Αφρική κυρίως είναι ε, η προέλευση και νέα όμως κράτη. Έχουμε νέες μεθόδους που χρησιμοποιούν διακινητές και λαθρέμπων ναρκωτικών και βάζουν την κοκαίνη σε πλαστικά, σε ιδιρουχισμού και έτσι την εισάγουν. Υπάρχουν εργαστήρια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, βρίσκονται δύο στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, όμως στην Πολωνία και τη Λιθουανία και αυτά καλύπτουν τις ανάγκες, τη ζήτηση αυτά τα ναρκωτικά. Βλέπουμε λοιπόν η παραγωγή να γίνεται όλο και πολύπλοκη για τα συνθετικά ναρκωτικά. Συχνά ε, χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες ε, μη ρυθμισμένες και η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα εξάγει έκσταση και αμφεταμίνες σε πολύ μεγάλο ε, βαθμό. Πρέπει να πω ολοκληρώνοντας ότι μπορούμε να αποκριθούμε σε εξελίξεις αυτές αποτελεσματικά εξελίξει που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά των ναρκωτικών, μόνο αν βασιστούμε σε καλά δεδομένα, πληροφορίες και σε ε, σωστή ανάλυση. Αυτό νομίζω ότι παρέχουμε με την έκθεσή μας το οργανωμένο έγκλημα, επενδύει σε νέα προϊόντα, σε νέε τεχνολογίε, σε νέε επιχειρησιακέ και λειτουργικέ πρακτικέ και προσεγγίσεις. Εμεί όμω συνεχίζουμε στην Ευρώπη να εργαζόμαστε για να εντοπίσουμε όλε τι νέε τάσει και για να ανταποκριθούμε ε, και προληπτικά. Η έκθεσή μα εστιάζει κυρίω στην αγορά ναρκωτικών. Πώ μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματικές δράσει. Βέβαια αυτό είναι μία από του νομίσματο. Η πρόοδο που θα πετύχουμε στο μέλλον θα βασιστεί στο αν μειωθεί και η προσφορά και η ζήτηση. Είναι κεντρική η προσέγγιση που θα έχουμε λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο σκελών τη προσφάση και τη ζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι η έκθεση για την αγορά των νοικοτικών είναι ένα καλό παράδειγμα που δείχνει ότι η κριτική και ψύχρεμη ανάλυση μπορεί να βοηθήσει. Χαίρομαι πολύ που το έκπνου του είχε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τη Europol για το πολύ σημαντικό αυτό project. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. We thank you. We thank you. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Γκιώτς για την παρουσίασή σας και για το έργο που κάνει το Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την ε, τοξικορμανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την Europol, τώρα και σου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση προς την Ευρωπόλη να παρουσιάσει την άποψή της σε αυτή την κοινή έκθεση και θέλω να πω και στον κύριο Γκέτς ότι ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή η συνεργασία μας με το δικό του φορέα. Αυτό δείχνει ότι αν μπορέσουμε να συνενώσουμε διάφορες αρμοδιότητες μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όπως ξέρετε η Ευρωπόλ είναι μια διοκτική υπηρεσία, βλέπει την πιο σκοτεινή πλευρά ε, του φαινομένου των ναρκωτικών. Ο κύριος Γκέτς βλέπει την πιο ορατή πλευρά κατά κάποιο τρόπο, αλλά από κοινού μπορούμε να καταλήξουμε σε πολλά αποτελέσματα. Έχουμε 1,4 εκατομμύρια παραπάνω ε, χρήστες μετά τον τελευταίο χρόνο και όπως είπε και ο κύριος Γκέτς περίπου 700 ακόμα ψυχοτρόπες ε, ουσίες έχουν εισαχθεί στην αγορά. Φοβάμαι ότι Παντού υπάρχουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχει χωριό, πόλη, κομμόπολη, ε, μεγάλη πόλη που δεν έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Τα αποτελέσματα είναι ληστείες, ε, διαρρήξεις, ε, φόνοι, εκβιασμοί που οφείλονται στους εμπόρους ναρκωτικών και επίσης πολλές φορές η εξάρτηση οδηγού πολλούς σε, στην εγκληματικότητα για να μπορέσουν να εξεύρουν τα προς, τα προς την πρέζαν τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν γνωρίζει ότι είναι πολύ μεγάλο το, το, το, το τμήμα των εγκλημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά, το μεγαλύτερο κομμάτι των εγκλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει αυτή η δραστηριότητα της διανομής ναρκωτικών μια βασική διαδικασία για τις εγκληματικές ομάδες. Δεν αντιμετωπίζουν μονάχα ένα είδος ναρκωτικών, αντιμετωπίζουν και ναρκωτικά και άλλες ουσίες, αλλά τα ναρκωτικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπορία αυτών των οργανώσεων αλλάζουν συνέχεια τους δρόμους λαθρεμπορίας και τους τρόπους με τους οποίους αποφεύγουν τη δίωξη. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν κάθε φορά να βρίσκουμε τρόπους να τους σταματάμε. Είδαμε να υπάρχει και μία αύξηση στην εξαγωγή ε, ναρκωτικών με νόμιμους τρόπους όπως είναι τα κοντέινερ, ταχυδρομικές υπηρεσίες, αεροπορικές πτήσεις είναι λοιπόν όλο και πιο δύσκολο να μπορέσει κανεί να διακριβώσει τι γίνεται. Δεν μπορεί να πάει σε ένα λιμάνι και να ελέγξει όλα τα κοντέινερ τα οποία μπαίνουν. Είναι αδύνατο να γίνει πλήρη έλεγχο όλων αυτών των αγαθών. Μία από τι πιο συνηθισμένε μεθόδου είναι η λεγομενη on λοιπόν rip-off. Ε, δηλαδή βασίζεται στην διαφθορά των υπαλλήλων στα λιμάνια <clears throat> με πολύ καλό συντορισμό των δραστηριοτήτων αυτών. Τα αγαθά στα κοντέινερ αντικαθιστώνται με λαθρέα αγαθά και επίσης το ίδιο πράγμα γίνεται και στον λιμένα προορισμού. Με τον τρόπο αυτό υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μπορούν να εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν τα ναρκωτικά. Η κοκαίνη όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Γκότς έρχεται κυρίως από την Νότια Αμερική και ε, διηλίζεται και εξευγενίζεται σε πολλές φορές σε χώρους στην Νότια Αφρική και μετά με κοντέινερ έρχεται στην Ευρώπη. Και το διαδίκτυο έχει παίξει σημαντικό ρόλο γιατί χρησιμοποιείται και τρόπος, ως τρόπος πώλησης ναρκωτικών. Τα πάντα μπορούν να αγοραστούν από το ίντερνετ. Πολλοί θεωρούν ότι είναι πιο εύκολο να αγοράσουν έτσι ναρκωτικά. Πολλές φορές μπορεί κανείς να το κάνει μέσω του ίντερνετ και μετά θα το ε, παραδώσει κάποιος όπως γίνεται και με τις πίτσες. Έχουμε λοιπόν αυτές τις αγορές τις επιγραμμικές που οδηγούν και σε μεγάλη μυστικότητα. Υπάρχουν ε, πολλές ε, διαδικασίες πληρωμής με ρευστά, με κάρτες πληρωμής και με άλλους τρόπους που είναι πολύ δύσκολο να ανοιχνευτούν αυτές οι πληρωμές. Αυτό είναι μια δυσκολία για τις διοκτικές δυνάμεις και πρέπει να είναι ένα από τα νέα στοιχεία στη νέα στρατηγική για το κυβερνοέγκλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Βλέπουμε ότι η κοκαίνη είναι το πρώτο ναρκωτικό στην Ευρώπη μετά την κάναβη. Οι εισαγωγέ κοκαίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίω οργανώνονται από εγκληματικέ οργανώσει εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια φιλελευθερωποίηση αυτή τη αγορά και πολλέ ε, οργανωμένε εγκληματικέ ομάδε μπορούν τώρα να προβαίνουν σε εισαγωγέ κοκαίνη στην Ευρώπη. Και το γεγονό ότι έχουν ε, εξαλειφθεί τα περισσότερα καρτέλ της Κολομβίας μετά από την προσπάθεια των Κολομβιανών και της DEA, της Αμερικανικής Υπηρεσίας για την Καταπλέμηση των Ναρκωτικών, φαίνεται ότι τώρα οι ευρωπαϊκές εγκληματικές ομάδες έχουν περισσότερες δοσοληψίες με τα καρτέλ του Μεξικού που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην διαμετακόμιση ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγού, παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν για να μπορέσουμε, όπως είπε και ο κύριος Μέτς, να ελαχιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα το αρνητικό της χρήση ναρκωτικών. Όχι μόνο η αστυνομία, οι μεταφορικέ υπηρεσίε, αλλά και οι άλλοι εμπλεκόμενοι, τα σχολεία, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνε και αθλητές που μπορούν να αποτελέσουν ε, υποδείγματα ρόλου, θα πρέπει να καταδείξουν ότι δεν είναι μαγιά το να χρησιμοποιεί κανεί ναρκωτικά και να αποτρέψουν του νέου από όλα από τη χρήση του. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκρέσ και την πολύ καλή συνεργασία και ελπίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι χρήσιμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ που μα προσκαλέσατε. Σα ευχαριστώ πολύ και του δύο. Έχουμε ε, τώρα και χρόνο για συζήτηση. Η κυρία Σίπελ θέλει το λόγο από ό,τι βλέπω και ενδέχεται και να ακολουθήσουν άλλοι από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ. Έχω ένα πάρα πολύ σύντομο ερώτημα. Αν κατάλαβα καλά αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Ευρωπόλ, είπε ότι τα αδικήματα που έχουν να κάνουν με ναρκωτικά από την ε, δράση των εγκληματικών οργανώσεων μέχρι τη δράση των απλών πρεζονίων αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των εγκληματικών πράξεων μέσα στην Ευρώπη. Γι' αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπόλ και οι εθνικές διοκτικές αρχές έχουν θέσει τα αδικήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά στο επίκεντρο των προσπαθειών τους και αν καταβάλουν τις μεγαλύτερες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τη μορφή εγκληματικότητας. Ευχαριστώ κύριε Αντωνέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές και καλεσμένους μας και θα ήθελα να αναφερθώ σε μία από τις πτυχές που αναφέρθηκε από τον κύριο Γκέτς στην παρουσίασή του. Τα λεγόμενα νόμιμα ναρκωτικά. Γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο, ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο που έχει αναδειθεί και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Έχει αυξηθεί η χρήση αυτών των νομίμων ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σοβαρότητα αυτού του φαινομένου έχει αναφερθεί προηγουμένως. Εγώ ε, έχω κάνει συζήτηση για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά έχει να πράξει πολύ περισσότερα σε σχέση με τον έλεγχο και την απαγόρευση πολλές φορές αυτών των λεγόμενων νομίμων ναρκωτικών. Γιατί τα λέμε νόμιμα καταρχήν. Είναι νόμιμα γιατί δεν έχουν απαγορευτεί. Δεν έχουν απαγορευτεί γιατί δεν είναι γνωστά. Γιατί η ταχύτητα της καινοτομίας για την αγορά αυτών των προϊόντων και η παγκοσμιοποίηση κάνουν το φαινόμενο αυτό πολύ δύσκολο να το ελέγξει κανείς. Από το 2010 η Κομισιόν μας έχει υποσχεθεί ότι θα προβεί σε μια αξιολόγηση των φαινομένων αυτών και θα καταλήξει σε κάποιες τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλέγμα το οποίο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση 307 του 2005 είναι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και προβλέπει κάποιους κάπως βαρύς και επαχθείς μηχανισμούς οι οποίοι είναι χρονοβόροι για να αντιμετωπιστούν οι ουσίες αυτές. Και θα σας δώσω κάποια στοιχεία από την έκθεση που συζητούμε σήμερα. Από το 1997 μόνο 12 ουσίες αξιολογήθηκαν από πλευράς ανάλυσης κινδύνου και απαγορεύτηκαν στην Ένωση. Όλοι συμφωνούν ότι μόνο με, ευρωπαϊκή, ε, με αντίθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό. Τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν μια σειρά εθνικών μέσων. Το γεγονός ωστόσο ότι τα, φάρμακα, τα ναρκωτικά αυτά πολλούνται στο ίντερνετ καθιστά αδύνατη, αδύνατο τον έλεγχο σε εθνικό πλαίσιο. Τώρα, πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. και πότε η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για νέο νομοθετικό εργαλείο που θα μπορούσε να προσφέρει μια λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Ευχαριστώ. Κύριε Χέρτ, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση πραγματικά υπάρχει μία ανησυχητική τάση για την αύξηση ε, των ναρκωτικών αυτών στους νέους που στρέφονται στα ναρκωτικά και όχι στο ενόπνευμα. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη αναφέρθηκαν. Πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει μια αναθεώρηση της οδηγίας για τα ναρκωτικά και να βρούμε μια λύση ως προς την ε, σχετική ευθύνη, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική. Λέγεται ότι, αναφέρθηκε ότι η Ευρώπη παράγει κυρίως συνθετικά ναρκωτικά. Όντως, υπάρχει ωστόσο κάποια εικόνα για το τι μπορεί να, γίνουν, ε, να γίνει στον τομέα αυτό. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση από πλευρά μα και να καταλάβουμε πώ μπορούμε να σταματήσει η παραγωγή αυτών των συμφερικών ναρκωτικών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλα, άλλες παρατηρήσεις, άρα ξαναστρεφόμαστε προ του δύο προσκεκλημένου μα. Κύριε Γκέτ, θέλετε να ξεκινήσετε ή κύριε Έτινγκ. Η η η πρωτη ερώτηση πήγαινε περισσότερο προ την αστυνομία, αν υπάρχουν ειδικευμένε μονάδες στα κράτη-μέλη και στη Europol. Σωστά είπε ο μιλητή, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που πρέπει να έχουμε ε, δεσμευμένη μονάδα για το σκοπό αυτό. Το τι συμβαίνει τώρα. Στις ανώτερε βαθμίδες του οργανωμένου εγκλήματος υπάρχει αλλαγή. Παλιά οι εγκληματίε. Κάποιοι ήταν καλοί στα χρηματοκιβώτια, άλλοι ήταν καλοί στις ληστείες, στις κλοπές. Τώρα είναι καλοί σε συγκεκριμένε δραστηριότητε, αλλά δεν ασχολούνται μόνο με συγκεκριμένε δραστηριότητε, ναρκωτικά για παράδειγμα. Οπότε τα περισσότερα κράτη στην Ευρώπη έχουν πιο ευέλικτε δομέ για να καλύψουν όλα τα, όλες τις ουσίες, τα, τα δικήματα που χρησιμοποιούνται. Βεβαίω έχουμε πάντα ειδικού για τα ναρκωτικά, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της παραγωγής των προδρόμων ανάλογα με την προέλευση και τους. Οπότε υπάρχουν ειδικέ μονάδες που έχουν ταυτόχρονα Έχουμε και ειδικευμένες μονάδες, έχουμε και συνολικές μονάδες που εξετάζουν τη, όλα τα προϊόντα κέρδη, ροή χρηματική, επενδύσεις τους. Δεν ξέρω αν αυτό απάντησε στην ερώτησή σας και μετά ο κ. Γκέτς θα απαντήσει. Οι άλλες δύο ερωτήσεις αφορούσαν και οι δύο τη, τα νομική διάσταση. Νόμιμη κλοπή. Το legal heist, ε, όπως αποκαλείται. Αυτό είναι περίεργος όρος, δηλαδή είτε είναι κάτι νόμιμο είτε όχι. Πάντως δεν, αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι νόμιμο. Αυτό που κάνει η Επιτροπή και, αυτό, και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει κυρίως η Επιτροπή είναι ότι ετοιμάζουν ένα νέο κείμενο για την αναδιατύπωση του κανονισμού του 2005 μετατρέποντας το σε ένα νέο νομικό εργαλείο βάσει της συναπόφασης. Αυτή τη στιγμή το σύστημα του 2005 λειτουργεί καλά, άρα έχει φτάσει στα ωριά του. Και το Συμβούλιο αποφάσισε ξεκίνησε την διαδικασία της νέας ουσίας που λέγεται 4MA και τώρα εξετάζει την ε, ε, τη νέα ουσία που λέγεται 4ET, 4ET. Και στις δύο περιπτώσεις η διαδικασία εξέτασης είναι θετική, αλλά τα προβλήματα της υφιστάμενης νομικής βάσης υπάρχουν. Δεν υπάρχει επαρκής ε, έλεγχος με την ε, δικαστική προσέγγιση. Ε, όταν συζητηθεί αυτό στην Επιτροπή σας θα σας ζητούσα να δείτε τι απαιτείται να προστεθεί στον κανονισμό για να προχωρήσει. Τώρα, τι μπορεί να γίνει για να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Είπα νωρίτερα, δεν μπορούμε να, γνω, να βλέπουμε κάθε ουσία χωριστά πλέον. Πρέπει να τις δούμε συνολικά. Είπε και ο συνάδελφος ότι πρέπει να βλέπουμε το οργανωμένο έγκλημα ευρύτερα με όλες τις, με όλες τις διαστάσεις ε, των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Και απλά θα σας έλεγα ότι τα εθνικά μέτρα δυστυχώς είναι απλώς ανεπαρκή. Μπορεί να είναι σκληρά, αλλά είναι ανεπαρκή. Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση ευρωπαϊκή στον τομέα αυτό. Αν δείτε τι προβλέπει η συνθήκη η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, η αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα των είναι εξαιρετικά ε, δυνατή και θα έπρεπε να δοθεί περαιτέρω ευρωπαϊκή διάσταση γιατί η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ε, είναι ευρωπαϊκή για να μην σας πω και παγκόσμια. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Όχι. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γκέτς και τον κύριο Έρτινγκ για την παρουσίαση της κοινή έκθεσης για την πανευρωπαϊκή αγορά ναρκωτικών. Αυτή την εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση για την ασφάλεια των πολιτών μας. Που εδώ ως αιρετοί τους εκπρόσωποι προστατεύουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, Το θέμα είναι γενικότερο διότι διαφορά και τον τροποποιητικό κανονισμό για τις ε, πρόδρομες ουσίες. Έχουμε την κυρία Χέντ εδώ, που θα συνεχίσει να μας παρουσιάζει τις, απόσ... τις απόψεις για τις πρόδομες ουσίες. Ευχαριστούμε τους προκεκλημένους μας. Ευχαριστούμε τους δύο εκπροσώπους ε, της ε, Europol που ήρθαν και μίλησαν και δίνω το λόγο στην κυρία Χέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα, ένα αρκετά τεχνικό θέμα οι πρόδρομοι είναι χημικέ ουσίε που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικέ μεθόδου για παραγωγή πλαστικών, φαρμακευτικών, καλλινικών αρωμάτων, απορριπαντικών, αλλά μπορούν συγχρόνω να χρησιμοποιηθούν και για παράνομε ναρκωτικέ ουσίε. Επομένως, υπάρχει ένα σύστημα αδειοδότησης και καταχώρησης για την παρακολούθηση της εμπορίας προδρόμων ουσιών. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε αντικείμενο κρατικής κριτικής συγγνώμη, για την αντιμετώπιση αυτών των ουσιών, για τον οξικό ανιδρύτη ιδίω, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παραγωγή τεχνητών ε, πλαστικών και τε, βαφών υφασμάτων κτλ. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί επωφελώς για την παραγωγή ηρωίνης, αμφεταμινών και κοκαίνης. Και πρόκειται ιδίως για την ηρωίνη. Είναι η βασική πρόδρομη για την ηρωίνη, η οποία ευθύνεται για πάρα πολλού θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση αυτή που παρουσιάστηκε προηγουμένω, δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην ε, εκτροπή του οξικού ανιδρύτη για την εγκληματική χρήση του για την παραγωγή ηρωίνης. Η πρόταση της Κομισιόν έχει σαν στόχο να περιορίσει το εύρος των ορισμών που χρησιμοποιούνται για τις ουσίες αυτές και να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση του εμπορίου του οξικού ανιδρύτη και να υπάρξουν πιο αυστηροί κανόνες για την καταχώρηση αυτού του αυτή τη διακίνηση και καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζουμε, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα αποτραπούν οι εγκληματικέ οργανώσει από το να χρησιμοποιούν την πιο, τον πιο ασθενή κρίκο μέσα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο επίση να δημιουργηθεί και μια τράπεζα δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα μπορέσει να διατηρήσει όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε μια καλύτερη επισκόψη για την κατάσταση τη ε, διακίνηση των προδρόμων ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ υποστηρίζω τι γενικέ γραμμέ τη Κομισιόν. Θεωρώ όμω ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο. Ιδίω σκέφτομαι για τα θέματα προστασία δεδομένων, όπου είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι η χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων θα υπόκειται σε σαφεί κανόνε και επίση αυτό αφορά ιδιαίτερα την χρήση τραπεζών δεδομένων. Επίση, ζητώ να παρακολουθηθεί πλήρως και η διαδικασία των, ε, της εμπορίας προδρόμων και η Κομισιόν μετά τρία χρόνια μετά τη θέση εφαρμογή της ε, οδηγίας αυτής να μας δώσει μία ε, έκθεση για να μας εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει η επισκόπηση αυτής της αγοράς. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα ήθελαν να μιλήσουν. Ακούσατε την παρουσίαση του σχεδίου έκθεση από την εισηγήτρια κυρία Χέντ. Δεν θέλετε να πείτε κάτι, μήπως θέλει να πει κάποιο άλλο θεσμικό όργανο, μήπως η Κομισιόν. Ο εκπρόσωπος Κλάους Μπέρεντ, ο εκπρόσωπος Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Χέντ για την έκθεσή της. Η, μάλιστα η έκθεση αυτή συντάχθηκε τάχιστα. Η Κομισιόν συμφωνεί με την πρόταση της ηγετρίας να εξασφαλίσει την κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι ένα θέμα που, του οποίου άπτονται πολλές από τις τροπολογίες. Σας στηρίζουμε την πρόταση. Όπως λέτε κι εσείς, στόχο έχει να αντιμετωπίσει τα ειδικά ε, χαρακτηριστικά του προβλήματος, ιδίως για τον οξικό ανιδρύτη. Στις τροπολογίες σας περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία κατά ω επιτοπλίστων μπορούμε να δεχθούμε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα είχαμε κάποια σχόλια παρόλα αυτά για θέματα που μας φαίνονται λίγο πιο πολύπλοκα, συγκεκριμένα. Νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή ασυνέπεια σε ό,τι αφορά τον περιορισμό, μάλλον το εύρος του περιορισμού των ευαίσθητων δεδομένων, μιλώ για την τροπολογία 6 και για την τροπολογία 14, όπου γίνεται αναφορά στο άρθρο 8 παράγραφο 1 τη Οδηγία 9546 Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Νομίζουμε ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή. Προτείνει η επίση επίσης να περιοριστεί η διατήρηση των αρχείων, μιλάω για την τροπολογία 7, μόνο δύο χρόνια. Και θα ήθελα να πω ότι ο υφιστάμενος κανονισμός προβλέπει διατήρηση των στοιχείων για τουλάχιστον τρία έτη. Αυτό δεν μας έχει δημιουργήσει στην πρακτική κάποιο πρόβλημα και υπάρχει κάποια σχέση με το εξωτερικό εμπόριο των πρόδρομων ουσιών. Και υπάρχει αυτή η ρύθμιση που προβλέπεται και από τον τελωνιακό κώδικα για τη διατήρηση των στοιχείων για τρία έτη και έτσι παραμένουμε συνεπείς και με άλλα σκέλη του κανονισμού για το εξωτερικό εμπόριο. Σε ό,τι αφορά 11, στις κατεξουσιοδότηση πράξη, καταλαβαίνουμε ότι λέτε πως θα πρέπει να αναφέρονται τα είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και είναι αντικείμενο επεξεργασία. Η μία μικρή δυσκολία που έχουμε με τη διατύπωση είναι εκεί που λέει κατόπιν έγκριση των κατεξουσιοδότη πράξεων, διότι η συλλογή για τις κατασχέσεις και για την αναστολή κάποιων αποστολών είναι στοιχεία τα οποία έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Θα έπρεπε λοιπόν αντί να λέτε κατέξι να λέτε σύμφωνα με. Δηλαδή το πρώτο βήμα έχει ήδη γίνει. Δεν υπάρχει συλλογή επεξεργασία ε, προσωπικών δεδομένων στο συγκεκριμένο στάδιο. Μιλάμε μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, για την κατάσχεση και την αναστολή ε, αποστόλων φορτίων. Τώρα, εκτιμούμε το γεγονό ότι σίγουρα πρέπει να επιβεβαιούται και η αποτελεσματικότητα των προτινόμενων κανονισμών. Λέμε εμείς ότι πρέπει να υπάρξουν πέντε χρόνια και μετά θα αναθεωρήσουμε, θα εξετάσουμε την πρόταση. Η συγκεκριμένη προτείνει τρία χρόνια. Εμείς γιατί προτείναμε πέντε χρόνια. Διότι στον εφιστάμενο κανονισμό υπήρχε μια τέτοια υποχρέωση αναθεώρηση μετά από τρία χρόνια, λέει ο, ο μιλητής. Και είχαμε συμφωνήσει ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα για να καταλάβουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικό ή όχι. Ουσιαστικά μετά από 1,5 χρόνο ξεκινούν οι έρευνε και οι διαβουλεύσεις για να έχουμε και την έκθεση σε τρία χρόνια. Προτείναμε λοιπόν σε συνεργασία με όλου του άλλου εμπλεκομένου η αξιολόγηση να γίνεται μετά από πέντε χρόνια. Για να έχουμε μπορέσει να δούμε τι επιπτώσει των ε, τροποποιημένων διατάξεων. Ουσιαστικά αυτά είχα να πω. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον πρόσωπο τη Κομισιόν, Ισλανδική Προεδρία. Μήπω πριν στρέψουμε πάλι στην εισηγητρία, την προσοχή μας. Άλλοι βουλευτές ενδεχομένως. Κύριε Πίρκερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι εξισορροπημένη αυτή η έκθεση, δεν δημιουργεί προβλήματα, αλλά έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις σχετικά. Η πρώτη παρατήρηση είναι η εξή. Αφορά και τα σημεία που ανέφερε και η Κομισιόν εκεί που η συγγήτρια προτείνει τα τρία χρόνια να γίνουν δύο για την ε, κράτηση των στοιχείων. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω γιατί και κατά πόσο αυτό συνδέεται με τις πρακτικές ε, συνέπειες. Νομίζω ότι τα τρία χρόνια είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε αποδεκτό γιατί ζητάει η συγγήτρια να γίνουν τα τρία χρόνια δύο. Θα ήθελα να μου το εξηγήσει. Και επίσης θα ήθελα να σταθώ στην τροπολογία 14 όπου αναφέρεται η χρήση πληροφοριών και της χρήσης τους μόνο για τους στόχους της, ε, του κανονισμού και να απαγορεύεται η διασύνδεση αυτών των ε, βάσεων δεδομένων με άλλες βάσεις δεδομένων. Μα είναι φανερό ότι αυτά τα στοιχεία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους στόχους αυτού του κανονισμού. Εγώ πιστεύω για αυτό το λόγο ότι αυτή η τροπολογία είναι περιττή, διότι δεν υπάρχει ένας ε, επακριβής ορισμός της χρήσης των στοιχείων που να προβλέπεται από αυτή την οδηγία. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι περιττή. Κατά τα άλλα, εγώ υποστηρίζω την ε, έκθεση της κυρίας Χέλη, η οποία νομίζω ότι έχει ένα πρακτικό χαρακτήρα και είναι απόλυτα εφαρμόσιμη. Ευχαριστώ. Κυρία Ρομέρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να θέσω ένα ερώτημα προς την ε, Εκτελεστική Επιτροπή για τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί εδώ από την εισηγήτρια σε σχέση με το ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη για τα προσωπικά στοιχεία. Καταρχήν ο επόπτης αυτός αφορά μονάχα στην, ε, στα στοιχεία που συνδέονται με τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όχι σε γενικότερο επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω το εξής ερώτημα στην Κομισιόν. Τι ρόλο πιστεύει ότι μπορεί να έχει εδώ ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων για το μητρό αυτό ή μάλλον αυτή τη βάση δεδομένων που αφορά τις ε, επιχειρήσεις και οι οποίες δεν είναι θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Επομένως είναι εκτός της σφαίρας εφαρμογής Το δεύτερο ερώτημα που ήθελα να θέσω είναι προς την Ευρωπόλ. Εφόσον η Ευρωπόλ είναι αρμόδια για τα σοβαρά εγκλήματα, θα ήθελα να ξέρω αν αυτά τα σοβαρά δικήματα που δεν έχουν να κάνουν βέβαια με την έκθεση HED αλλά με, έχουν μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν η Ευρωπόλ θεωρεί ως σοβαρά εγκλήματα αυτά τα οποία αναφέρονται και στην Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Δηλαδή τα 32 αυτά δικήματα που αναφέρονται σε αυτή την νομοθετική πράξη. Δεν βλέπω κανέναν να θέλει το λόγο να πω απλά ότι δυστυχώς έχοντας ακούσει τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ναρκωτικών στην Λισαβόνα και της Europol και χωρίς άλλες παρεμβάσεις πέρασαμε στο επόμενο σημείο την έκθεση της κυρίας Χέντ. Έφυγαν εν τω μεταξύ και οι εκπρόσωποι από την Υπηρεσία Ναρκωτικών και την Europol πάντω. Αν θέλετε μπορεί να στείλετε την ερώτησή σας μέσω της Επιτροπής μας. Εγγράφος ή να περιμένετε να έρθουν την άλλη φορά που θα έρθουν αυτοί. Εδώ. Τέθηκε ωστόσο και μια συγκεκριμένη ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της ε, επιτροπή. Δεν ξέρω αν κύριε Μπέρεντ μπορείτε να απαντήσετε πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια εκ Ευχαριστώ. Να απαντήσω και σε αυτό που είπε ο κύριος Πίρκερ για την τροπολογία 14. Ξέχασα να το πω στην πρώτη μου παρέμβαση. Καταλαβαίνω την επιμήγεια της εισηγήτριας να υπάρξει σαφής περιορισμός ως προς το στόχο της χρήσης των δεδομένων. Πιστεύω ωστόσο ότι αν είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί από ό,τι προτείνεται εδώ θα ήταν κάτι χρήσιμο. Τα στοιχεία Φερρυπίν για τους εμπλεκόμενους σε ύποπτες συναλλαγές θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη διάλυση οργανωμένων δικτύων ε, διακίνησης ναρκωτικών. Αν λέμε μόνο στην πρόληψη των της ε, εκτροπής προδρόμων ουσιών θα χάναμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες για άλλα άτομα που εμπλέκονται σε δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών. Τώρα, για το ρόλο του, του Ευρωπαϊκού Επιόπτη Προστασίας Δεδομένων, του EDPS, η κυρία Ντορομέρο σωστά αναφέρει ότι τα περισσότερα συλλογικά δεδομένα, ε, ε, προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και την χάνουν επεξεργασίας ε, βρίσκονται σε, γίνονται σε επίπεδο κρατών μελών πρώτα και μετά μπαίνουν στις ευρωπαϊκές βάσεις. Αν κατάλαβα καλά ωστόσο, η εισηγήτρια στην έκθεσή της περιλαμβάνει και κάποιες τοπολογίες που θα διευκρινίζουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των εθνικών ε, δομών προστασίας δεδομένων και ζητείται να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και του Ευρωπαϊκού έλεγκτη προσωπικών δεδομένων. Η δική μας εμπλοκή ποια είναι. Πρώτον, ζητήσαμε την γνωμοδότηση του EDPS, πήραμε την γνωμοδότηση λεπτομεριακή και νομίζω ότι ο εισηγητής υιοθετεί πολλές από τις παρατηρήσεις ε, της έκθεσης του EDPS στις, τροπολογίες, στις τροπολογίες της. Μία τροπολογία μάλιστα λέει ότι όλες οι κατεξοδότησεις πράξεις που υιοθετούνται για το είδο των προσωπικών δεδομένων που θα αποθηκεύονται, αν αποθηκεύονται στην ευρωπαϊκή βάση, θα πρέπει να έχουν και την γνωμοδότηση του EDPS. Θα το κάνουμε. Θα υπάρχει μια σχετική διαβούλευση. Επίσης, σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση που πρέπει να δίνεται στον, στο υποκείμενο των δεδομένων για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες διόρθωσης τυχών ε, εσφαλμένων πληροφοριών. Σίγουρα θα εμπλακεί ο EDPS σε κάθε φάση των δραστηριοτήτων μας στην ε, διαχείριση και λειτουργία των, ε, της βάσης δεδομένων. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου πρόεδρος. Κυρία Χέντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <coughs> Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στη συζήτηση. Θα λάβω υπόψη τις απόψεις που διατύπωσαν. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την εργασία μας. Υπάρχει τώρα ένα ερώτημα το οποίο τέθησε μένα για την τροπολογία υπαριθμών 7 για την ε, διατήρηση για δύο για τρία χρόνια των προσωπικών στοιχείων. Εδώ υπάρχει η σύμβαση του ΟΗΕ η οποία προβλέπει τέτοιου είδου στοιχεία να διατηρούνται μόνο για δύο χρόνια. Και δεν υπάρχει κανένας αποχρόν λόγος για να διατηρήσουμε τα στοιχεία αυτά για τρία χρόνια. Γι' αυτό έχω καταθέσει αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις ε, τροπολογίες και την ψήφιση αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα να ακούσω από τα χείλη του εισηγητή, του Προέδρου, συγγνώμη η προθεσμοί για τις τροπολογίες προτείνεται να είναι στις 28 Φεβρουαρίου, φέτος βέβαια, του 2013, το μεσημέρι. Και στη συνέχεια το επόμενο στάδιο της διαδικασίας θα ακολουθήσει. Υπάρχει ένα σχόλιο ακόμα για την Ευρωπόλη θα έχουμε μια ακρόαση του εκτελεστικού διευθυντή της ε, Ευρωπόλ, του Roth Ράιτ. προβλέπεται στις 21 Μαρτίου να λάβει χώρα, δηλαδή 23, 21 Μαρτίου λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε ερωτήματα στον κύριο Ράιτ σε σχέση με τα σοβαρά αντικείμενα και το ρόλο της Ευρωπόλ στα πλαίσια αυτά. Ναι. Οπότε είχαμε συμφωνήσει να αλλάξουμε την ε, σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να έχουμε την έκθεση της κυρίας Μακοβέη για την κατάσχεση στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες δεν είναι παρούσα η κυρία Μακοβέη, οπότε πρέπει να κάνουμε διάλειμμα ο λίγων λεπτών, δηλαδή μισή ώρα. Ευχαριστώ.

Ναι. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Σ' ακούω, αλλά πολύ χαμηλά σ' ακούω. Ένα, δύο. Μια χαρά σ' So, Mrs. McAvey not here. Λοιπόν, η κυρία Μακοβέη είναι εδώ. Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Το πηγαδάκι στο βάθος μπορούν οι συνάδελφοι αν θέλουν να καθίσουν για να ξανασυνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Κυρία Μακοβέη, Είναι το δικό σας θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τώρα την εργασία μας μετά από μια διακοπή λίγων λεπτών. Είμαστε στο σημείο υπαριθμών 9, το οποίο άλλαξε χρονική αλληλουχία. Πάγωμα και δίμευση των ε, προϊόντων εγκληματικών ενεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μακοβέη λοιπόν είναι αρμόδια εισηγήτρια για το θέμα αυτό. the change of the agenda. Now we are discussing the compromise amendments on the report on confiscation. Okay. Let's Ας συζητήσουμε για τις τροπολογίες συμβασμού και θα δώσω το λόγο στην κυρία Μακοβέη και μετά... Έχετε το λόγο κύριε Μακοβέη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως θυμόσαστε, έχουμε συζητήσει τις τροπολογίες Θα ήθελα να πληροφορήσω την Επιτροπή μας ότι έχω ήδη συναντηθεί με τους κοιόδης εισηγητές. Έχουμε συμφωνήσει για ορισμένες τροπολογίες συμβιβασμού σε μια ιδιαίτερα καρποφόρα συζήτηση γιατί υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις, πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις μεταξύ των κρατών μελών για τα θέματα αυτά και αποκλίνουν οι θέσεις των διαφορετικών κρατών μελών. Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία πάντως των εισηγητών συμφωνεί, των σχεδόν εισηγητών συμφωνεί σε ορισμένα σημεία. Επειδή πολλές τροπολογίες είχαν κατατεθεί επί τη βάση των εθνικών νομοθεσιών που όπως είπα προηγουμένως είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Προσπάθησα να καταλήξω καλή την σε συμβαστικές λύσεις οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους. Και θέλω να ευχαριστήσω τους και οδησυγητές για την υποστήριξή τους προς τις τροπολογίες συμβιβασμού αν χρειάζεται τώρα να συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες, είμαι απόλυτα διαθέσιμη να προβώ σε συζήτηση. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν να αναφερθούν στις τροπολογίες συμβιβασμού μετά από τη συζήτηση με τους κοιόδης εισηγητές. Και πάλι είμαι πολύ ευτυχισμένη για αυτά που έχουν γίνει και μέτρη να ακούσω τι απόψει των συναδέλφων. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Υπάρχει κάποιο που θέλει να λάβει το λόγο. Η κυρία Βέβα έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είμαι Μεταξύ αυτών που είχαν ζητήσει συζήτηση σήμερα για τις συμβασικές τροπολογίες, διότι διαβάζοντας τις ε, συνειδητοποίησα ότι ορισμένα από αυτά που περιλαμβάνουν δεν εφηγραμμίζονται καθόλου με αυτά που περίμενα εγώ. Και ένας άλλος λόγος είναι γιατί λάβαμε την ε, νομική εκτίμηση, την ε, νομοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου που γύρει κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φιλοσοφία ε, της δίμευσης δέσμευσης αλλά και με την νομική βάση της ε, εν λόγω οδηγίας. Τι μπορεί να περιλαμβάνεται και τι όχι δηλαδή. Λυπούμε γιατί ξέρω ότι ήταν πολύ καλή συνεργασία της εισηγητρίας με ορισμένου σκιώδης, μεταξύ αυτών και με το σκιώδη από την Άλντε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η άποψη του Σκιώδους είναι μεμονωμένη, απομονωμένος στην ε, ομάδα μας σχεδόν. Ο, ο Σκιώδης το συζητήσαμε και χθε και από ό,τι προέκυψε ξεκάθαρα είναι μια άποψη που δεν συμμερίζεται άλλος παρά μόνο η Σκιώδης της ομάδας μου. Φυσικά και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να σκοτώσουμε, αν με επιτρέπετε την έκθεση, την έκθεση αυτή. Το αντίθετο και ακριβώς γι' αυτό θέλαμε να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τροποποιήσεις εκεί που θεωρούμε ότι δεν είναι ε, παραδεκτές είτε από νομικής απόψεως είτε από πλευράς περιεχομένου αυτές τροπολογίες. Ιδάλλω στην αυριανή ψηφοφορία θα υπάρχουν λίγες ψήφοι υπέρ μόνο και περισσότερε περισσότερες θα είναι αρνητικές. Και αυτό γιατί βλέπω να εκφράζονται παρόμοιε αποψίσεις και από τους πρασίνους αλλά και από κάποια μέλη του ΕΛΚ. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι πολλά μέλη ε, και από το ομάδα των σοσιαλιστών, δημοκρατών ε, θα μας υποστηρίξουν. Τώρα έρχομαι στα πιο συγκεκριμένα. Από νομικής πλευράς νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε την ανάλυση της νομικής μας υπηρεσίας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι μεν η οδηγία αυτή εδράζεται επί μιας νομικής βάσης που ε, απτεται της, ε, συνεργασίας, ε, της συνεργασίας σε ποινικά ζητήματα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο που θα ρυθμίσουμε τα αστικά, τις αστικές υποθέσεις. Δηλαδή να επιβάλλουμε τα κατώτερα πρότυπα τα οποία προβλέπουν τι αστικέ υποθέσει, χωρί όμω να επηρεάσουμε τα ανθρώπινα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν είναι αυτό ο τρόπο αντιμετώπιση με την δέσμευση και την ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Άρα από αυτή την πλευρά. Θέλω να καταλάβω τη θέση τη εισηγήτρια. Δηλαδή, βιάζεται η εισηγήτρια, ε, πρέπει να ψηφίσουμε αύριο. Και αν ναι, γιατί. Γιατί τόση βιασύνη, γιατί τόση σπουδή. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ψηφίσουμε αύριο. Είναι πιο χαλαρό το θέμα. Νομίζω μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πρώτα μεταξύ μα Οι διάφορε πολιτικέ ομάδε. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ και εγώ κυρία Βέμπερ. Ο κύριο Ντε Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τη Μόνικα Μακοβέη για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Καταρχήν, είμαι υπέρ των συμβαστικών τροπολογιών. Στην πλειονότητά τους, με εξαίρεση δύο. Θα ανέφερα προς το τέλος η κυρία Μακοβέη. Νομίζω το ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει εδώ είναι η ανεπίσημη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας που λάβαμε. Νομίζω ότι στην ουσία της λέει αυτή η νορμοδότηση ότι στο ποινικό δίκαιο οι απαιτήσει για ε, αποδεκτικά στοιχεία είναι υψηλότερες σε σχέση με το αστικό δίκαιο. Και αυτό είναι μια αφετηρία ε, αιτιολογημένη. Αλλά Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται για να καταδικαστεί κάποιος για ένα αδίκημα οι αρχές ισχύουν, αλλά είναι διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνουν τι συμβαστικέ τροπολογίε. Εδώ όμω δεν μιλάμε για καταδίκη, για κάποια εγκληματική πράξη, αλλά μιλάμε για δίμευση. Και μιλάμε για τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται ώστε να αποδείξει κανείς ότι προς ε, κατάσχεση, δίμευση, περιουσία έχει να κάνει κάτι με ε, το έγκλημα, με μια εγκληματική δραστηριότητα έμεσα ή άμεσα. Προσωπικά λοιπόν πιστεύω ότι οι συμβιβαστικές τροπολογίες της Μόνικα, τις οποίες κατάρτισε συνεργασία με τους και ηγητές, μπορούν να παραμείνουν ως έχουν, όμως, και εδώ θα συμφωνήσω με την Βέμπερ, ότι πρέπει να δούμε πάρα πολύ προσεκτικά τα πράγματα και νομίζω ότι αυτό πιο πολύ θέλω να πω. Επειδή έχουμε τα ποινικά ζητήματα εδώ, ε, πρέπει να έχουμε χρόνο για να σκεφτούμε με ηρεμία και ψυχραιμία. Δεν ξέρω αν θα έχουμε αρκετό χρόνο σήμερα στη συζήτηση να επισέλθουμε σε αρκετό βάθος και για να εξετάσουμε και τα επιχειρήματα της γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε περισσότερο χρόνο για αυτή τη συζήτηση. Θέλω πάντως να ξεκαθαρίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαι ακόμη πεπισμένος ότι η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας θα πρέπει να επηρεάσει τι βασικέ τροπολογίε κατά κάποιο τρόπο. Θα ήθελα πάντω να έχω χρόνο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε καλύτερα και με ε, περισσότερο χρόνο και με την νομική υπηρεσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι συμβαστικέ τροπολογίε, έχω κάποιε παρατηρήσει για την υπαριθμόν 3, για το τι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ε, διήμευση. Νόμιζα ότι το κείμενο ήταν αρχικά ισορροπημένο. Εξαιρούνταν δηλαδή από τις δημεύσεις, από τη δίμευση αγαθά που είναι απαραίτητα προς το ζήν. και τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν έναν πλήρη κατάλογο όλων αυτών των αγαθών. Εγώ θα είχα να διατυπώσω ε, μια ε, εναλλακτική πρόταση. Παραμένω στη δική μου ε, πρόταση τροπολογία και δεν θέλω να υποστηρίξω την τρία Ούτε και τη δέκα συμβιβαστική τη βρίσκω σωστή, γιατί ουσιαστικά υπαγορεύει στα κράτη-μέλη τι θα κάνουν. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει άλλος άμεσα διαθέσιμο προορισμό, οι πρόσοδοι από τα ε, αποκλιματικέ δραστηριότητε θα χρησιμοποιούνται για σκοπό τη πρόληψη εγκληματικών Δεν νομίζω ότι αυτό όμως είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τις δημεύσει στην Ευρώπη. Το τι κάνουν τα κράτη-μέλη με τις προσόδους των δημεύσεων ε, δεν μας ε, αφορά. Στο παρόν πλαίσιο τουλάχιστον. Νομίζω ότι πιο πολύ προέκυψε από το ιταλικό παράδειγμα. Συμφωνώ με τη Ρενάτε Βέμπερ, αλλά θέλω να πω στην Άλντε ότι στην πρώτη συζήτηση που είχαμε εδώ σε επίπεδο επιτροπής ο εκπρόσωπος της Άλντε είχα προσέξει ότι είχε ήδη τότε πει και μιλήσει για κάποια ζητήματα που και εγώ δεν αναγνώριζα ως γενική άποψη της ομάδας Άλντε. Και θα ήταν πολύ καλύτερο για την εισηγήτρια και για τους κοιόδης εισηγητές αν η άλλη είχε καταλήξει ε, σε μια κοινή άποψη στην αρχή και όχι στο τέλος. Κυρία Σίπελ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά δεν εκπροσωπώ την άποψη πολιτικής μου ομάδος αυτή τη στιγμή με αυτά που σας λέω, αλλά μπορώ να σας πω ότι έχω δυσκολίες για να υποστηρίξω αυτή την έκθεση. Στις συμβαστικέ τροπολογίες υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία για μένα είναι ιδιαίτερα προβληματικά. Πάντα έχουμε ένα πρόβλημα με την ε, ανάμειξη του αστικού δικαίου με το διοικητικό δικαίου, δικαίου, θα πρέπει τα θέματα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε πιο προσεκτικά. Το θέμα των αρμοδίων αρχών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ελέγξουμε ιδιαίτερα προσεκτικά και επίσης το ερώτημα του με ποιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία τα οποία είναι στη διάθεσή μας προτού πώς θα αξιογίνει η αξιοποίηση αυτών των στοιχείων προτού προβούμε σε μια δίμευση ή δέσμευση. Το άρθρο 10 μου φαίνεται προβληματικό, δηλαδή το ότι τα κράτη τα οποία κάνουν αυτήν την ε, δέσμευση μπορούν να διερευνούν ποιος ε, είναι ο αποδέκτης, ποιος θα, καρπεί, θα καρπούτο αυτά τα ποσά όταν δεν υπάρχει μια ποινική δίωξη εναντίον τους που να έχει κινήσει. Όλα αυτά με κάνουν να είμαι πολύ διστακτική για να δεχτώ αυτή τη συμβαστική λύση. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ. Είχα αναφέρει και προηγουμένως την δική μου θέση και είχα τονίσει ότι για ορισμένα λεπτομεριακά σημεία της έκθεσης έχω μεγάλα προβλήματα. Και δεν πρόκειται μονάχα για πολιτικά προβλήματα, αλλά είναι και προβλήματα νομικής φύσεως, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό θέλω να επιμείνω. Όσοι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, οι κανόνες που έχουν να κάνουν με το δίκαιο της ιδιοκτησίας αποτελούν πραγματικά μια απειλή για τα νομικά συστήματα των χωρών μας. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητος, υπάρχει το δίκαιο στην ιδιοκτησία, υπάρχει το βάρος ε, απόδειξης το οποίο δεν μπορεί να αναστραφεί στις ποινικέ υποθέσεις. Εδώ βλέπουμε τον κίνδυνο να υπάρξει μια αυθαίρετη νομική ρύθμιση βάσει αυτής της ε, οδηγίας. Αυτό δεν μπορεί λοιπόν να συμβεί και εγώ Έχω ζητήσει να υπάρξει και κάποια επαλήθευση άτυπα από τις νομικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι όλες αυτές οι, οι αντιρρήσεις και οι ανησυχίες που έχω μπορεί εσείς να μην τις πάρετε στα σοβαρά όταν προέρχονται από μένα προσωπικά, αλλά όταν υπάρχουν αμφιβολίες και από τη νομική υπηρεσία δεν μπορείτε να τις παραγνωρίσετε και δεν μπορείτε ελαφρά την καρδία να αποφασίσετε για θέματα ουσίας χωρίς να λάβετε υπόψη αυτές τις νομικές πτυχές παραδείγματος χάρη στην ε, τροπολογία συμβιβασμού 9. Όταν λέμε ότι κάποιος δεν είναι σε θέση να αποδείξει την νόμιμη προέλευση ορισμένων αγαθών, αυτό είναι αναστροφή του βάρους απόδειξης. Αυτό δεν είναι αυτό το οποίο ήθιστε να ισχύει ένα κράτος δικαίου. Με όλη την καλή θέληση που έχουμε, με όλη την προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε να εμποδίσουμε τους εγκληματίες να αποκτούν αγαθά από εγκληματικές δια, ε, διαδικασίες, δεν μπορούμε εμείς να υπάρχει ένας αποχρόν λόγος να ανατρέψουμε το ισχύο νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά το βάρος απόδειξης. Θα πρέπει να παραμείνουμε λοιπόν μέσα στα πλαίσια τα οποία θεσπίζει το εθνικό δίκαιο των χωρών μας για τις ποινικέ διαδικασίες και να προσαρμόσουμε έτσι τις τροπολογίες συμβιβασμού στο ισχύον δίκαιο. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι απαραίτητο για μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μην γίνουμε, ε, ώστε να μην γελιοποιηθούμε ουσιαστικά και να δείξουμε ότι δεν σεβόμαστε τις έννοιες του δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Λάτφορντ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με όσους θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε αύριο δεδομένου ότι φαίνεται να υπάρχουν ε, πολλά ουσιαστικά προβλήματα στο κείμενο. Δεν, είμαι, δεν ήμουν βέβαια σκιώδης, αλλά ανησυχώ με ένα ιδιαίτερο θέμα που αναφέρθηκε από τον κύριο Καϊόλα, τον ε, νομικό σύμβουλό μας. και με οδήγησε στο να κάνω μια σειρά απολογιών, ιδίω στην 94. Δεν βλέπω στις του απολογίε της κυρίας Μακοβέη να αντικατοπτρίζονται οι θέσει μας. Η οδηγία αυτή βασίζεται στα άρθρα 82 και 83, δηλαδή οι νομικές βάσεις που σχετίζονται με τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής, ε, του ποινικού δικαίου. Εισάγει δηλαδή εισάγει ωστόσο μέτρα αστικής δικονομίας μέσω της οδηγίας. Ορισμένα κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων είμαι ξεκάθαρη είναι και η Βρετανία ήδη έχουν μέτρα διατάξεις στο αστικό δίκαιο που επιτρέπουν τη δυνατότητα κατάσχεσης χωρίς ποινική καταδίκη. Όπως είπε η κυρία Μακοβέη, αυτό θεωρήθηκε ότι το, δικαστήριο, το, το, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι τούτο συμβαδίζει με την ΕΣΔΑ. Η ιδέα είναι να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη που έχουν τώρα συστήματα κατάσχεσης δια του αστικού δικαίου να κρατήσουν τα συστήματα αυτά. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τούτο είναι εκτός πεδίου εφαρμογής οδηγίες. Δεν είναι η διατύπωση της κυρίας ε, Μακοβέη που λέει ότι τούτο δεν, ε, ότι οι διατάξεις αυτές είναι με την επιφύλαξη των εθνικών ρυθμίσεων που επιτρέπουν κατάσχεση ε, βάση αστικού δικαίου. Αυτό δημιουργεί μια φαιά που δεν καθιστά σαφές το νομικό πλαίσιο, σε δύο κράτη τουλάχιστον. Όταν υπάρχει κατάσχεση βασιαστικού δικαίου, τα δύο κράτη-μέλη που υπάρχουν μπορούν μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν με τον τρόπο χωρίς να χρειάζονται ρυθμίσεις ποινικού δικαίου. Δηλαδή, συνεχίζουν να διατηρούνται οι δυνατότητες κατάσχεσης ή δίμευσης που προϋπήρχαν χωρίς την ενσωμάτωση της οδηγίας. Αυτό είναι μια σημαντική διάκριση. Και δεν είμαι βέβαιη ότι θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν καταλαβαίνω και δεν συμφωνώ επίσης με μια άλλη πρόταση στο email του κυρίου Καϊόλα ότι όταν υπάρχει δυνατότητα κατάσχεσης βάσει του αστικού δικαίου, οι κανόνες που εφαρμόζονται εκεί δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερης ποιότητας από τους κανόνες που εισάγει η οδηγία. Εγώ αν κατάλαβα καλά από την προηγούμενη παρέμβαση του ήταν ότι συμφωνούσε πως η οδηγία αυτή δεν μπορεί να εισάγει εξουσία αστικής κατάσχεσης, ότι απλά μπορούν να συνεχιστούν οι υφιστάμενες, ε, ε, ε, οι υφιστάμενες ρυθμίσεις. Η ανησυχία μου σε κάθε περίπτωση με την πρόταση κ. Μακοβέ είναι ότι παρουσιάζει, ότι εισάγει μάλλον, έλλειψη ασφάλεια δικαίου για το πεδίο εφαρμογή οδηγίε, που εγώ προσπαθώ, αν καταλαβαίνω καλά, αφορά αποκλειστικά ποινικέ ρυθμίσει. Ο κ. Κίρκοπ. Συμφωνώ με τις προγενέστερες παρατηρήσεις. Εδώ γίνεται μνήμα στα ένομα συστήματα, το οποίο λειτουργεί στον πληθυντικό. Δηλαδή έχουν πολλές ε, ρυθμίσεις και πολλά συστήματα δικαίου που επιτρέπουν ή όχι την κατάσχεση βάσει ποινικών ε, αποφάσεων. Εμένα με ανησυχεί η καθυστέρηση που θα πετύχει απλά μια συνένεση δεν οδηγεί πουθενά, διότι δεν μπορεί να πετύχουμε συνένεση όταν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από κράτο σε κράτο. Κάποια ευρωπαϊκά κράτη, και εγώ εδώ υποστηρίζω την κυρία Μακοβέη στι προσπάθειε τη να προχωρήσουμε, υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν το θέμα της δίμευση των ε, προϊόντων του εγκλήματος δια της αστικής οδού. Προφανώς ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος θέλει τα παράνομα κέρδη παράνομη συμπεριφορά... να μένουν στα χέρια εγκληματιών ή συνεργών τους. Από Βρετανική στη Βρετανία τσεκάραμε το θέμα αυτό από την οπτική γωνία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το επιχείρημα ότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι πιστικό πλέον. Βεβαίως, πρόεδρε, ορισμένες χώρες κατέστησαν σαφές ότι δεν μπορείς να δημεύσεις, να δημεύσεις τα στοιχεία αυτά εκτός αν έχεις μία απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σοβα... Ε, ουσιαστική καταδίκη ενός ατόμου. Αυτό το καταλαβαίνω. Σημαίνει, μάλλον αυτό σημαίνει ότι όσοι μιλούν από αυτή την οπτική γωνία χρησιμοποιούν τη δική τους εμπειρία και μπορεί να τη δικαιολογήσουν. Το βασικό θέμα, πρόεδρε, ωστόσο, είναι να έχουμε επαρκές περιθώριο ούτω ώστε οι χώρες οι οποίες λειτουργούν διαδικασία δίμευσης με, με, ασφάλι, με, ασφαλιστικές δικλείδες διά της αστικής οδού να μπορούν να τις συνεχίσουν να το κάνουν. Τώρα, αν κάποιες χώρες θέλουν να χρησιμοποιούν και την ποινική διαδικασία, σημαίνει ότι μπορούμε συνολικά, σαν Ένωση, να, κατασ... να... να... να δημεύουμε τις περισσότερες, ε, τα περισσότερα προϊόντα του εγκλήματος. Αυτό το υποστηρίζω. Επίσης υποστηρίζω αυτό που είπε η Λέβη Λάτφορντ. Δεν μπορούμε να κλείσουμε την δυνατότητα αυτή. Θα ήταν παράλογο και εξαιρετικά επικίνδυνο να προχωρήσουμε μέσω της οδηγίας στην διακοπή του δικαιώματος να ασκούμε τη δυνατότητα να δεσμεύουμε διατιαστικής οδού ό,τι αφορά ε, προϊόντα εγκλήματος. Κυρία Ματιέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας κάποιους από τους συναδέλφους προηγήθηκαν διερωτώ με μήπως τελικά δεν έχουμε συζητήσει επαρκώς το κείμενο μεταξύ μας. Το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά αυτό που έχουμε μπροστά μας σήμερα δεν το έχουμε συζητήσει αρκετά. Γι' αυτό και προκύπτουν ε, ορισμένα προβλήματα και οι συνάδελφοι εκτιμούν ότι υπάρχουν προβλήματα με τα θεμελιώδη δικαιώματα, με ορισμένα από τα συντάγματα, των κρατών νομικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Τώρα τι πρέπει να γίνει δεν ξέρω, αύριο λογικά πρέπει να ψηφίσουμε, αλλά τίθεται το ερώτημα αν έτσι όπως έχουν τα πράγματα και όπως έχει το κείμενο, αν πράγματι ε, είναι σκόπο να ψηφίσουμε αύριο ή όχι. Τώρα σε ό,τι αφορά την ε, νομοδότηση της νομικής υπηρεσίας, τι να σας πω, εμείς πρέπει να πάρουμε την απόφαση, αλλά και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε μάλλον να εξετάσουμε τον ενδεχόμενο να αναβάλουμε την ψηφοφορία και το θέτω στη Μόνικα. Να το σκεφτεί. Να έχουμε δηλαδή πρώτα κάποιες συναντήσεις και να το συζητήσουμε ξανά γιατί δεν με έχει ικανοποιήσει ούτε και η σημερινή συζήτηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Μακοβέη. Κυρία Μακοβέη. Ακούσατε τα σχόλια ορισμένων συναδέλφων. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ξέχασα την κυρία Μπορσελίνο. Συγγνώμη. Είχα ζητήσει το λόγο νωρίτερα και δεν ήθελα να σε διακόψω. Καταρχάς θέλω να υπενθυμίσω ότι μιλούμε για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και ευαίσθητο μιλούμε για την δέσμευση ή δίμευση προϊόντων εγκλήματος που είναι πάμπολα. Ξέρουμε τα νούμερα. Παρότι δεν είναι οριστικά και σαφή τα στοιχεία, αλλά σίγουρα μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για εγκλήματα, σοβαρότατα εγκλήματα που πρέπει να ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουν όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παιδική πορνογραφία, εμπορία ανθρώπων, ε, σεξουαλική εκμετάλλευση, ε, εγκληματικότητα που συνδέεται με τα ναρκωτικά. Είναι ένα πολύ λεπτό ευαίσθητο θέμα και πιστεύω ότι η συζήτηση έτσι όπως διατυπώνεται δείχνει ακριβώς την προσοχή που δίνουμε σε αυτά τα θέματα. Εργαστήκαμε καλά με την κυρία Μαρκοβέη, συζητήσαμε επί μακρόν, προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις όλων και τη σκέψη όλων των συναδέλφων που δούλεψαν για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι οι συμβαστικές τροπολογίες που είναι οι πλέον συζητήσιμες αφορούν την δέσμευση, την, την δίμευση χωρίς καταδίκη και τον αποδέκτη. Και άρα αυτό είναι δείγμα ότι στο στη νομική διάσταση ε, επικεντρώνουμε την προσοχή μας, όπου νομίζω ότι υπάρχει και εκτεταμένη συμφωνία. Εγώ θα... Ε, αναφέρθηκε και η προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας θυμίζω ότι και το ΕΔΑΔ έλαβε θετική θέση για διαδικασίες που χωρίς ε, ποινική καταδίκη σε περίπτωση επικινδύνων, ατόμων επικινδύνων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια επιτρέπουν την δέσμευση προϊόντων. Δεν υπάρχει λοιπόν βλάβη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα τουλάχιστον με την ομολογία του Στρασβούργου. Κατόπιν, να υπογραμμίσω και κάτι ακόμα. Έχω μια προσωπική εντύπωση, παράξενη και το λέω προσωπική εντύπωση γιατί είμαι σκιώδης για τους σοσιαλιστές. Την ομάδα θα τη δω μόνο στη μία σήμερα, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος της ομάδας. Προσωπικά σχολιάζω. Θέλω απλά να υπογραμμίσω ότι μίλησε ο συνάδελφος Γιόγκ για τα ουσιώδη αγαθά που δεν μπορούμε να τα ε, δεσμεύσουμε παρότι τα πήρε ε, παράνομα. Αυτό θα έπρεπε να μας οδηγήσει να σκεφτούμε ότι τα αγαθά που απέκτησε ο εγκληματίας τα απέκτησε από κάποιον άλλον. Το να μιλάμε λοιπόν για την προστασία των ουσιωδών αγαθών ενός ανθρώπου που ε, ζει, πάντων που εμπλέκεται σε τέτοια αδικήματα πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη σε δεύτερο επίπεδο, αφού προστατεύσουμε τα δικαιώματα πρώτα του ατόμου που αρχικά ευλάβηκαν. Τα άτομα δεν είναι τα επιμέρους τα, θύματα, δεν είναι τα άτομα τα θύματα, αλλά η κοινότητα, ε, το θύμα της οργανωμένης εγκληματικότητας είναι η κοινωνία κατά βάση, στο σύνολό της. Από αυτή την οπτική πρέπει να δούμε την κατάσταση, διαφυλάσσοντας το θύμα, την κοινωνία δηλαδή. Είδαμε προηγουμένως ε, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήδη η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλύπτεται. Αλλά μέσα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να προστατεύουμε και το θύμα του εγκλήματος. Πιστεύω ότι Πρέπει όχι μόνο να προσέχουμε ιδιαίτερα το τι γράφουμε και το τι συζητούμε. Πρέπει ταυτόχρονα να δώσουμε τη δέουσα προσοχή και σε αυτό το μήνυμα που θα περάσουμε στην κοινή γνώμη. Το να είμαστε τόσο διαιρεμένοι σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα σίγουρα θα δώσει αρνητική ε, εντύπωση. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ψηφιστούν οι διατάξεις αυτές και να δούμε ποια είναι η λύση προσπαθώντας να προσεγγίσουμε όσο περισσότερο γίνεται τις θέσεις μας όπως έγινε και θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλά να ψηφίσουμε ούτως ή άλλως δεν είναι οριστική ψηφοφορία. Ένα βήμα είναι στην πορεία που θα μας οδηγήσει στην οριστική ψηφοφορία. Πιστεύω ότι μία αναβολή θα έδινε αρνητική εικόνα δίνοντας δηλαδή την εντύπωση ότι το κοινοβούλιο είναι διαιρεμένο και ευαίσθητο ζήτημα. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες. Θέλω να μιλήσω με την ομάδα μου πρώτα, αλλά θέλω να σας δώσω αυτή τη γενική προσέγγιση μου και τον τρόπο που θα πρέπει να προχωρήσουμε. Κατά άποψή μου είναι σημαντικό και το μήνυμα που δίνουμε προς τα έξω δεν πρέπει να είναι ένα μήνυμα κοινοβουλίου που χωρίζεται, που διαιρείται, αλλά που προσανατολίζεται στο βασικό στόχο, την προστασία της κοινωνίας και των δικαιωμάτων της, τη, ε, ε, διώκοντας, κυνηγώντα τόσο σοβαρά αδικήματα. Η κυρία Βέμπερ θέλει να κάνει κάποια σχόλια, παρακαλώ σύντομα. Καταλαβαίνω αυτά που είπε η κυρία Μπορσελίνο όταν αναφέρεται στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας και των εγκληματιών και των διαφόρων κατηγοριών. Κοιτάξτε όμως την τροπολογία συμβιβασμού υπαριθμών 9. Δεν υπάρχει τίποτα για τη συγκεκριμένη αξιόπινη εγκληματική πράξη. Απλώς λέει ότι αν κάποιος δεν μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευση των στοιχείων των αγαθών, των στοιχείων ενεργητικού που έχει. Μα αυτή είναι η νομοθεσία που είδα εγώ στη δική μου χώρα και μπορώ να σας πω το επίπεδο αυθαιρεσίας που προέγυψε ξεπερνάει κάθε μορφή φαντασίας. Θέλουμε κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Μακοβέη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με την νομική βάση. Θέλω να κάνω το εξή σχόλιο. Είμαι ίδια νομομαθής και δικηγόρος. Και έχω φέρει και θέματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι ήταν η 20η υπόθεση που έφερα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο ΕΔΑΔ και την κέρδισα και αυτήν πριν από δύο εβδομάδες. Γνωρίζω λοιπόν την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και σας έχουμε στείλει σε όλους τις σχετικές ε, αποφάσεις του δικαστηρίου. Αυτό συνδέεται και με τη νομική βάση. Η δίμευση εμπίπτει στο άρθρο 83 ανεξάρτητα από το αν θεωρείται ε, ποινή ή απλώς διοικητικό μέτρο και βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο για τις ε, ποινικέ κυρώσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικές δραστηριότητες το πάγωμα και η δίμευση των περιουσιακών αγαθών σε περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας. Όλες οι τροπολογίες λοιπόν βρίσκονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μιλάμε για ένα άλλο πλαίσιο το οποίο εκφεύγει των δράσεων του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Πράγματι λοιπόν, είναι ένα μέτρο αντιμετώπισης των εγκληματικών ενεργειών και είναι κάτι που συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διαβάστε τα email σας. Σας έχω στείλει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά. Και πάλι, μιλάμε για δίμευση που δεν βασίζεται σε απόφαση καταδικαστική. Και σας το ξαναλέω. Ακόμα και αν χρησιμοποιείτε αυτό σε αστικές υποθέσεις δεν αντιμετωπίζεται ως ε, θέμα αστικής δικαιοσύνης γιατί συνδέεται πάντα με, τη δραστηριότητα, με κάποια δραστηριότητα εγκληματικού χαρακτήρα. Δεν θα σχολιάσω απόψεις όπως γιατί πάμε βεβαιασμένα σε μια ψηφοφορία ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό το είχαμε αποφασίσει να ψηφίσουμε όλοι μαζί για αύριο. Και νιώθω έκπληξη αυτή τη στιγμή που χθες άρχισαν να έρχονται email ζητήσανε συζήτηση για τις ε, συμβαστικές τροπολογίες έγινε αυτή η συζήτηση χρειάζεται όμως καλύτερος συντονισμός αν εγώ καλή την πίστη συζητώ με όλους τους σκιώδεις εισηγητές και καταλήγουμε σε μια συμφωνία για τις συμβιβαστικές τροπολογίες, έχω κάθε λόγο να ελπίζω ότι αν όχι η απόλυτη πλειοψηφία όλων, αλλά τουλάχιστον μια πλειοψηφία υποστηρίζει αυτήν την ε, θέση. Έχουμε ακόμα κάποιες διαφωνίες, θα ξανασυζητήσουμε το απόγευμα αλλά εναπόκειται σε εμά να δούμε πώς θα μπορέσουμε μέσα στι ομάδε μας να δούμε αν υπάρχει ή όχι μια πλειοψηφία. Μπορούμε να μην ψηφίσουμε σημαντικέ λύσει και να ψηφίσουμε κάθε παράγραφο χωριστά. Αλλά δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Είχαμε ήδη αποφασίσει να κάνουμε την ψηφοφορία αύριο. Συμφωνώ όμω ότι για να έχουμε μια περαιτέρω συζήτηση και διευκρίνηση για αυτού που χρειάζονται διευκρίνηση, εγώ δεν χρειάζομαι περαιτέρω διευκρίνηση, μπορώ να αναβάλω την ψηφοφορία, να δεχτώ την αναβολή της ψηφοφορίας για τον επόμενο μήνα, αν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο. Και διαβάστε, σα λέω και πάλι, τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε περίπτωση δίμευση, χωρί να υπάρχει βάση καταδικαστικής απόφασης. Το ότι αυτό συνάδει λοιπόν με την ομολογία του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με τη Σύμβαση για τα Ανθρωπίνα Δικαιώματα. Μάλιστα, μας έχετε στείλει ένα email και το μήνυμα που λαμβάνουμε τώρα είναι ότι προτείνεται αναβολή Τη ψηφοφορία. Βέβαια αυτό πρέπει να το αποφασίσει η Επιτροπή μας γιατί η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί όπως γνωρίζετε για αύριο, για την 21η Φεβρουαρίου. Εάν θέλετε αναβολή πρέπει να το αποφασίσουμε τώρα. Ποιε είναι οι θέσει των εκπροσώπων των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Συμφωνείτε να αναβάλουμε αντιρρήσει. Yes, yes, I see, I see, I see. Βλέπω ότι το ΕΛΚ συμφωνεί. Οι φιλελεύθεροι συμφωνούν. Οι σοσιαλιστές δεν έχουν ένσταση. Οι πράσινοι τι πρεσβεύουν. Τα βάρες. Συμφωνούμε με την αναβολή. Αλλά θα ήθελα να κάνω μία πρόταση. Πρώτα απ' όλα, αν συμφωνεί η γήτρια, θα ήθελα να προτείνω να ζητήσουμε την επίσημη τοποθέτηση της νομικής υπηρεσίας, γιατί νομίζω ότι οι συντονιστές πρέπει να το ρωτήσουν, αλλά Αν συμφωνήσει η γήτρια. Πρόεδρος. Κύριε Μπορσελίνο. Μπορώ να συμφωνήσω για την αναβολή εφόσον η αναβολή αυτή δεν ε, παρατείνεται μακρόν για τους λόγους αυτούς που εξήγησε στην προηγούμενη παρέμβασή μου. Φυσικά και δεν είναι επάδοστον η αναβολή. Θα ψηφίσουμε απλά στην μεθεπόμενη επίσημη συνεδρία της ομάδας μας, δηλαδή το Μάρτιο θα ψηφίσουμε. Μιλάμε για το πολύ ένα μήνα δηλαδή αναβολή. Υπάρχουν σχόλια από την κυρία Μακοβέη. Πριν και δώσω στο λόγο να δώσω λόγο στον κύριο Κύρκοπ. Ο κύριος Κύρκοπ. Κύριε Πρόεδρε, Μπορώ να παραχωρήσω αυτή την αναβολή μόνο όμως αν ο προτραχικός στόχος της αναβολής είναι για παράδειγμα να ζητήσουμε περαιτέρω καθοδήγηση και από την νομική υπηρεσία για τα σημεία τα οποία ετέθησαν και από τις δύο πλευρές. Αν όμως αυτό γίνεται απλά και μόνο για να έχουμε μεγαλύτερο, ε, περισσότερο χρόνο στη θέση μας για να καταλήξουμε σε συνένεση, ε, όπως είπα και στην προηγούμενη παρέμβασή μου, υπάρχουν ε, κάποιοι δύσκολοι τομείς στα διάφορα νομικά συστήματα που δεν μπορούν απλά έτσι να τα ξεκαθαρίσουμε τόσο απλά. Μόνο λοιπόν για το λόγο που σας προανέφερα θα δεχθώ την αναβολή. Πρόεδρος, ακούσαμε λοιπόν ε, την υπόδειξη να μας ξεκαθαρίσει τα νομικά η νομική υπηρεσία. Πάντως από ό,τι φαίνεται συμφωνείτε όλοι να αναβάλουμε την ψηφοφορία για ένα μηνάρι. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τον Μάρτιο. Ε, να απόκειται τώρα σε εσά. Κυρία Μακοβέως, ιδιαίτερα να πείτε την τελευταία κουβέντα. So yes, in March. Ωραία. <clears throat> για την νομική βάση, όπως είπα προηγουμένως, όπως ανέφερα και άλλες δύο φορές προηγουμένως, βλέπω ποια είναι η νομική βάση, είμαι νομομαθής, σας έχω στείλει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ξέρουμε τη συνθήκη. Δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση από την νομική υπηρεσία, για μένα τα πράγματα είναι κρυστάλλινα σαφή. Έχει σταλεί ένα email από τη γραμματεία, ανεπίσημα, εντάξει. Για μένα τα πράγματα είναι σαφή. Εγώ είμαι έτοιμη να σας ε, εξηγήσω και πάλι και να συζητήσω με τους χειώδεις εισηγητές τι ισχύει για την νομική βάση. Γιατί η νομική υπηρεσία ήταν παρούσα σε ώρες της συνεδριάσης μας, όπως γίνεται πάντα. Θα ήθελα να ζητήσω και από τη Γραμματεία λοιπόν να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών αφού συζητήσουν προηγουμένως με τις πολιτικές ομάδες. Προτείνουμε, ε, εφόσον συμφωνείτε, να γίνει η επόμενη συνάντηση το Μάρτιο. Εσείς λέτε ότι δεν χρειάζεται νομική διευκρίνηση. Εσείς θεωρείτε τα πράγματα είναι σαφή, δεν ξέρω. Αν έχουμε μια συμφωνία λοιπόν για την αναβολή. Κυρία Λάτφορντ. Εγώ συμφωνώ για την αναβολή βέβαια, <clears throat> αλλά μπορώ να σας δώσω μονάχα τη δική μου οπτική γωνία. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια νομική γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία. Για μένα ο τρόπος με τον οποίο έχει διατυπώσει τις, νομικές, τις ε, συμβαστικές τροπολογίες η κυρία Μακοβέη δημιουργεί πολλές αμφιβολίες για το αν έχει καταλάβει αυτά που είπε νομική υπηρεσία. Ε, νομίζω ότι υπάρχει και μια γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου που μπορεί να πάρει η δική μα νομική υπηρεσία και θα ήταν χρήσιμο να πληροφορηθούμε κατά πόσο συμφωνούν οι δύο νομικέ υπηρεσίε. Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τις διακρίσεις που πρέπει να ισχύουν και τις δυνατότητες να ρυθμιστούν θέματα ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό το θέμα θα ανακύψει και σε άλλα νομοθετήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια σαφήνεια για το θέμα αυτό. Και φοβάμαι ότι διαφέρω με, σε επίπεδο άποψης με την κυρία Μακοβέη. Δεν θέλω να διαφυσβητήσω την γνώμη της και τη γνώση της, αλλά δεν είμαι σίγουροι ότι όταν συνέταξε τροπολογία 9, ότι έχει λάβει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Ωραία. Βλέπω να υπάρχουν πολλά μέλη τα οποία επιμένουν στο να υπάρξει προσφυγή στις νομικές υπηρεσίες Κύριε Ταβάρες. Θέλετε το λόγο. Με την ευκαιρία αυτή θα έλεγα να το συζητήσω και με τους συντονιστές πρώτα πρώτα πριν να αποφασίσουμε. Όχι. Προτείνω να αποφασίσουμε τώρα. Κύριε Ντε Είναι σημαντική, σημαντικό να έχουμε μια επίσημη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας γιατί αλλιώς ως συντονιστές ε, κάνουμε συζητήσεις νομικών θεμάτων και μετά αφού κάνουμε τις συζητήσεις λέμε καλύτερα να ακούσουμε ε, τους νομικούς. Καλύτερα το ξεκινήσουμε από τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία για να ζητήσουμε την άποψη της ε, ε νομικής και η S&D συμφωνεί και η ECR, η GUE, η Πράσινη, η Ωραία. Θα ακούσουμε την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και θα ψηφίσουμε τον Μάρτιο. Βεβαίως, επαναλαμβάνω όπως είπα, είμαι δικηγόρος, μελέτησα, σπούδασα, έχω άποψη για την νομική βάση. Αν κάποιοι χρειάζονται τη νομική υπηρεσία να τους βοηθήσει, να το συζητήσουμε. Η νομική υπηρεσία δεν αντικαθιστά τους συζητητές. Ωραία, το καταλάβαμε και σα έστειλα τα δίκτυα αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ωραία. Αυτό. Έχουμε και άλλο θέμα Τη κύρια Μακοβέη. Κατάσταση, ναι. Έχουμε ένα άλλο θέμα με την ίδια εισηγήτρια, την κυρία Μακοβέη. Αλλά θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Κόρκοραν, επικεφαλής του γραφείου του Ιρλανδικού Γραφείου Ανάκτησης ε, των ε, Προϊόντων του Σερβίου μας. Είναι εδώ ο κύριος Κόρκοραν. Παρακαλώ κύριε Κόρκοραν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κόρκοραν, Ευγένιο Κόρκοραν με λέμε. Είμαι υπεύθυνο ε, του Γραφείου ανάκτησης ε, των προϊόντων ποινικών ε, πράξεων στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία έχει μια σειρά σχετικά ανεπτυγμένων ε, νομικών δυνατοτήτων ανάκτησης προϊόντων εγκλήματος χωρίς καταδίκη δια της αστικής οδού. Στην παρουσίαση που θα σας κάνω σήμερα προτείνω να σας δώσω μια εικόνα της υπηρεσία μου αλλά και του νομικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί. Θα προσπαθήσω δεν να απαντήσω και σε ερωτήσεις που μπορεί να προκύπτουν ε, μπορεί να προκύπτουν από αυτό. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι εγκληματίες στην Ιρλανδία είχαν τη δυνατότητα να αυτοπροστατευτούν από ποινικά, ποινική δίωξη και σταδιακά οργανωμένοι εγκληματίες προστατευόταν χωρίς, επειδή δεν εμπλέκοντο ε, ευθέως σε κάποιες ποινικέ πράξεις και για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μορφή οργανωμένου εγκλήματος, λήφθηκαν μια σειρά μέτρων για να στερήσουν τους εγκληματίες αυτούς από την απόλαυση των ε, προϊόντων του εγκλήματός τους. Εισάγαμε λοιπόν ε, μορφές δέσμευσης ε, των προϊόντων, των κερδών από τα εγκλήματα για ε, για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά το 1994. Με μια, ο νόμος αυτός περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεων και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στην ποινική δίωξη. Σύντομα, ωστόσο, σε ένα χρόνο, στην πραγματικότητα, χρειαστήκε ακόμα πιο φιλόδοξο σύστημα για να αντιμετωπίσουμε τη διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα μετά την ε, δολοφονία ενός δημοσιογράφου που έκανε σχετική έρευνα και ενός ε, αστυνομικού σε υπηρεσία. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει δύο νόμους. Την, το νόμο θέσπισης του γραφείου μου και το νόμο για τα προϊόντα εγκλήματος την ίδια χρονιά, το 1995, που ήταν ε, η βάση της δέσμευση, του καθεστώτος δέσμευσης των προϊόντων εγκλήματος χωρίς ποινική καταδίκη στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία λειτουργήσε καλά, πέτυχε, είχαμε τη δυνατότητα να χτυπήσουμε μια σειρά εγκληματικών οργανώσεων με βάση αυτήν την νομοθεσία. Το ίδιο το νομοθετικό κείμενο αντιμετώπισε μια σειρά στιβαρών προκλήσεων τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω τι έπαθαν, τι, τι, τι αντιμετωπίσαμε. Το 1996 ενσωματώθηκαν, έγιναν μια σειρά, όπως σας είπα, νομοθετικών αλλαγών, ιδιαίτερα το μοντέλο δέσμευσης χωρίς ποινική δίωξη βάσει της, της προ, προαναφερθήσεως νομοθεσίας. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε μια πολυεπιστημονική προσέγγιση με ευθύνη στοχοθέτηση των προϊόντων και όχι του εγκλήματος, προϊόντων και όχι το ίδιο το έγκλημα. Χρησιμοποιούσαμε φερρυπίν το φορολογικό, τον κώδικα φορολογίας για τη δέσμευση των προϊόντων αυτών. Επίση, εισήχθησαν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που επιτρέπουν την ε, παροχή πληροφοριών ε, εμπιστευτικού χαρακτήρα μεταξύ των διαφόρων ε, νομικρατικών φορέων. Η υπηρεσία μου περιλαμβάνει αστυνομικούς, εφοριακούς, τελωνιακούς, υπαλλήλου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, νομικούς και διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Η δύναμη του γραφείου μας είναι η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας ως συνέχεια, ξεπερνώντας τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές υπηρεσίες. Η συνεργασία επιτυγχάνεται για της νομοθεσίας που επιτρέπει την αποκάλυψη συγκεκριμένων ε, εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων δομών των κρατικών υπηρεσιών που επιδιώκουν τους νόμιμους στόχους. Όπως σας είπα, στο γραφείο μου έχουμε δικηγόρους και λογιστές που δουλεύουν μαζί. Και αυτό κατά τη διάρκεια των ετών διαπιστώσαμε ότι έχει πολλά θετικά στοιχεία, επιτρέποντας καλή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού. Η διαθεσιμότητα της άμεσης παροχής πληροφοριών όλων των ειδών μέσα στο γραφείο είναι εξαιρετικά θετική επίσης. Ε, είναι αυτόνομος φορέας, αλλά ο επικεφαλής σύμφωνα με την νομοθεσία είναι αστυνομικό. Επιθεωρητής και άνω. Είναι υπόλογος στον αστυνομικό διευθυντή για την ε, λειτουργία, ενώ επιπλέον υπάρχει και ένα επιπλέον επίπεδο λογοδοσίας, μια και η υπηρεσία μας παρέχει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στον Υπουργό Δικαιοσύνη που το παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο μας. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το δημόσιο. Δεν έχει προκαθορισμένους οικονομικούς στόχους και τα έσοδα πηγαίνουν επίσης στο κρατικό προπολογισμό. Κάποιοι από τους στόχους ε, του, της υπηρεσίας είναι να χρησιμοποιήσει όλες τις δυναμικές δυνατότητες που έχει το κράτος για να διώξει σοβαρά, σοβαρά εγκρήματα. Κατά βάση χρησιμοποιούμε την νομοθεσία του 96 για τα προϊόντα εγκλήματος που προανέφερα. Χρησιμοποιούμε τον ποινικό κώδικα τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και τον κώδικα κοινωνικής ασφάλισης. Τα κέρδη των ε, προϊόντων εκμήματος φορολογούνται και η υπηρεσία μας έχει δυνατότητα, ευρύες δυνατότητες έρευνας και δέσμευσης. Πριν ε, πριν δημιουργηθεί το γραφείο μας υπήρχε μικρότερη βούληση των, ε, φορο, εφοριακών να κάνουν τέτοιες δεσμεύσει γιατί φοβόντουσαν για την ασφάλειά τους. Η παρουσία μας ενίσχυσε τη δυνατότητα των ε, υπαλλήλων των ε, φορολογικών υπηρεσιών να προχωρούν σε δεσμεύσεις, ε, μια και υπάρχει και η πολιτική και η οικονομική υποστήριξη. Ταυτόχρονα. Δεν έδειξαν μεγάλη, ε, μεγάλο δισταγμό στο να μειώσουν κοινωνικές παροχές και να αντιμετωπίσουν υπερβολικές πληρωμές σε σχέση με αυτούς που είχαν προσποριστεί εισοδήματα από το έγκλημα. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζει αρχές του αστικού δικαίου στα, στις προσόδους από εγκλήματα. Αν μπορεί λοιπόν το γραφείο μας να πείσει ένα δικαστήριο επί τη βάση πιθανοτικών συλλογισμών ότι τα αγαθά αυτά είναι προϊόν εγκλήματος, μπορεί να υπάρξει πάγωμα αυτών των αγαθών. Αυτή η απόφαση του δικαστηρίου ισχύει για 21 μέρες ε, κατά τη διάρκεια των οποίων το γραφείο μας ζητάει να γίνει μια διαδικασία για πιο μακροχρόνιο πάγωμα. Η αίτηση αυτή γίνεται και έναντι οποιοδήποτε ο οποίος έχει κάποιο ενδιαφέρον για αυτά τα αγαθά. Εάν λοιπόν διατηρηθεί, εάν γίνει αυτό, διατηρείται αυτό το πάγωμα μέχρι, από, μέχρι την πλήρη απόφαση του δικαστηρίου. Αν το δικαστήριο εκτιμήσει ότι στην πλήρη ακρόαση αυτά τα αγαθά είναι προϊόν εγκληματικής ενέργειας, μπορεί να υπάρξει μια μακροχρόνια ε, διαδικασία παγώματος για 7 χρόνια το λιγότερο. Μέσα σε αυτό το, διάστημα, εάν κάποιος μπορεί να πει στο δικαστήριο ότι τα αγαθά αυτά δεν είναι αποτέλεσμα εγκλήματος, μπορεί να εξασφαλίσει την άρση την ακύρωση αυτής της απόφασης. Εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία σε αγαθά που είναι τουλάχιστον αξίας 13.000 ευρώ που εκπροσωπούν το προϊόν του εγκλήματος. Επίσης η νομοθεσία δίδει, προβλέπει και τη δυνατότητα να, δώσουν, να δοθούν οι εκτιμήσεις ε, αρμοδίων αστυνομικών αρχών ή αρμοδίων φορολογικής αρχής ότι πράγματι τα στοιχεία αυτά ε, ενεργητικού είναι πράγματι άμεσα ή έμεσα προϊόν εγκλήματος. Η νομοθεσία και η εφαρμογή της νομοθεσίας έχει και υπόκειται και σε διασταυρούμενους ελέγχους για να μην υπάρξουν αδικίες. Η βασική δικλίδα ασφαλείας προβλέπει ένα σύστημα νομικής αρρωγής για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να υπομισθούν το κόστος των διαδικασιών. Το γεγονός ότι όλες αυτές οι δράσεις του γραφείου μας υπόκειται σε έλεγχο από τα δικαστήρια και ότι η ρήτρα για την ε, χρήση στοιχείων που αποτελούν μονάχα πεπιθήσεις και αυτή υπόκειται σε νομικό έλεγχο. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την πεποίθηση, μπορεί να ανατραπεί. Το γεγονός λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει δίμευση αυτής της περιουσίας είναι το, η τελική απόλυξη αυτής της διαδικασίας. Έχει υπάρξει και νομική διαμφισβήτηση αυτού του νομοθετήματος και έχουν αναφερθεί πολλά συνταγματικά επιχειρήματα τα οποία αντανακλούν ε, <clears throat> επιχειρήματα που αρίονται της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα αυτά έχουν έλθει ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας και μερικά από τα πιο σημαντικά επιχειρήματα τα οποία αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν το γεγονός ότι η ίδια η νομοθετική πράξη παραβίαζε το Ιρλανδικό Σύνταγμα γιατί ουσιαστικά δημιουργούσε μια ποινική διαδικασία με άλλο όνομα και επίσης το ότι η αστική διαδικασία δεν εξασφαλίζει τις δικονομικές ε, ε, διασφαλίσεις που προβλέπονται όπως παραγωγός το τεκμήριο αθωότητος και η απόδειξη της ενοχής πέραν λογικής αμφιβολίας. Με βάση αυτών των ε, επιχειρημάτων αποφάσισε το ανώτατο δικαστήριο ότι η κατάσχεση αγωθών είναι αστικό μέτρο και όχι ποινικό μέτρο και το δικαστήριο δεν έχει το δικαίωμα να διατάξει την κράτηση ή τη φυλάκιση οποιοδήποτε ατόμου και επίσης δεν υπάρχει καμία διαδικασία που να προβλέπει τη φυλάκιση ενός ατόμου εάν δεν ε, καταβάλει το πρόσημο το οποίο προβλέπεται. Επομένως θεώρησε τώρα το δικαστήριο ότι αυτές οι διαδικασίες δεν συγκροτούν ποινική διαδικασία. Το συμπέρασμα του του δικαστηρίου λοιπόν είναι ότι η κατάσχεση αυτή δεν είναι ποινική ποινικό κολασμός και οι διαδικασίες αυτές δεν αποτελούν ποινικέ διαδικασίες. Ένα δεύτερο επιχείρημα το οποίο ετέθη για να διαμφισβητηθεί αυτό το νομοθέτημα είναι ότι αυτή η πράξη αποτελεί, η νομοθετική πράξη αποτελεί αναστροφή του βάρους αποδείξεως. Το ανώτατο δικαστήριο θεώρησε ότι αυτή η αναστροφή λειτουργεί μόνο εάν είναι ικανοποιημένο το δικαστήριο ότι ορισμένα θέματα έχουν τεκμηριωθεί και υπάρχει απόλυτα πεποίθηση του δικαστηρίο ότι άμεσα ή έμεσα τα αγαθά αυτά είναι, είναι αποτέλεσμα ε, εγκληματικών ενεργειών. Υπάρχει επίσης δυνατότητα να υπάρξει αντεξέταση των μαρτύρων από το γραφείο και άλλες υπηρεσίες και υπάρχει και η δυνατότητα να ε, Διαμφισβητήσει κάνει το γεγονός ότι διεπράχθη κάποια εγκληματική ενέργεια για την απόκτηση αυτών των αγαθών. Το τελευταίο επιχείρημα το οποίο αναφέρθηκε είναι ότι αυτό το νομοθέτημα παραβιάζει την συνταγματική διάταξη κατά της αυτοενοχοποίησης και το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να εξισωθεί με μια συνταγματική επιταγή που αναγκάζει κάποιο άτομο να δώσει στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι αυτοενοχοποιητικού χαρακτήρα. Έχει αποφασιστεί λοιπόν με την ομολογία του ανώτατου δικαστηρίου ότι το κράτος μπορεί να παίξει και κάποιο ρόλο για την ε, δίμευση αυτών των αγαθών και η ιεραρχία ε, αγαθών δεν μπορεί να ερμηνευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε το ιδιωτικό δικαίωμα στην ιδιοκτησία μπορεί να υπερκεράσει το δημόσιο δικαίωμα κατάσχεσης. Η πράξη αυτή λοιπόν εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατάσχεση αγαθών από ιδιώτες, από μεμονωμένα άτομα, αλλά αναφέρει ότι αυτοί οι οποίοι έχουν αγαθά βάσει εγκληματικών δικαστηρίων δεν έχουν δικαίωμα σε αυτή την ιδιοκτησία την οποία απέκτησαν με παράνομα μέσα. Για παράδειγμα, δύο περιπτώσεις που αντιμετώπισε το γραφείο μας στην Ιρλανδία στο πρόσφατο παρελθόν και καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και, και το πώς ε, έχει εφαρμοστεί η διαδικασία αυτή για σχετικά ίσονες υποθέσεις. Μια τέτοια περίπτωση ξεκίνησε από εμάς μαζί με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ του 2010 και του 2012 και ο κύριος στόχος αυτής της ενέργειας αφορούσε ένα άτομο το οποίο είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε χρησιμοποιήσει τα προϊόντα αυτής της εγκληματικής ενέργειας για να αγοράσει ιδιοκτησίες στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης καταθέσεις σε τράπεζες και ένα τμήμα αυτών των εσόδων επενδύθηκε στην Ιρλανδία. Και υπήρξε συνεργασία των αστυνομικών αρχών και των ε, φορολογικών αρχών των δύο χωρών μαζί με το γραφείο μας. Τα έσοδα αυτά, οι πρόσοδοι αυτοί, έχουν επενδυθεί εν μέρη προωθεί για 100.000 μονάχα ευρώ για την αγορά δύο έγκυων ιδιοκτησιών στην Ιρλανδία και χρησιμοποιήθηκαν επίσης περαιτέρω πρόσοδα, πρόσοδοι για να ε, εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει αυτές τις ιδιοκτησίες και να τις χρησιμοποιήσει μαζί με μια εταιρεία αξιοποίησης. Λόγω της ε, ανόδου των ε, τιμών ιδιοκτησίας στην Ιρλανδία υπήρξαν σημαντικά κέρδη τα οποία προσπορίστηκε ο ενδιαφερομένος και υπήρξαν σημαντικά τα κέρδη που αποκόμισε από την πώληση αυτών των αγαθών που ήταν στην κατηγορία των ε, ιδιοκτησιών που αγοράζει κανείς και ξαναπουλάει αμέσως μέσα ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να εκμεταλλευτεί την άνοδο της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή πήρε ο εγκληματίας δάνεια της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ χρησιμοποιώντας ως ενέχειρο τις, ε, τις ιδιοκτησίες αυτές. Και μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο να, με διάφορους ενδιάμεσους να αποστασιοποιηθεί από τα αγαθά αυτά και χρησιμοποίησε τα χρήματα τα οποία κέρδισε για να αγοράσει άλλες ιδιοκτησίες. Χάρη στην άνοδο της αγοράς μπόρεσε να αποκομίσει όλο και περισσότερα χρήματα και να τα μεταφέρει σε τραπεζικούς λογαριασμούς <clears throat> στο όνομά του. Στο τέλος της ε, διαδικασίας αυτής, της κοινή έρευνας, το γραφείο μα κατάφερε να ανακτήσει 2,7 εκατομμύρια από τραπεζικούς λογαριασμούς, μεταξύ των οποίων 500.000 από αξιόγραφα που είχε στην Ιρλανδία το άτομο αυτό. Συγχρόνως καταδικάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι τώρα φυλακισμένος εκεί. Όπως σας είπα, ανακτήσαμε περίπου 3 εκατομμύρια από το άτομο αυτό. Ένα δεύτερο παράδειγμα μιας τέτοιας ενέργειας, η οποία έγινε στην Ιρλανδία, ήταν η λεγόμενη επιχείρηση Αλόχα. Κύριε να, κύριε να σας παρακαλώ, λέει. Ναι. Έχουμε χρόνο μόνο μέχρι τις 12.30 και έχουμε και άλλα σημεία στην μέση διάταξη. Αν μπορείτε όμως να συνοψίσετε γιατί έχουμε και άλλα θέματα και υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν. Αν μπορείτε να καταλήξετε. Να πω απλώς, λέει ο κ. Κόρκαραν, ότι η κατάσχεση χωρίς δικαστική απόφαση είναι κάτι το οποίο έχουν θεωρήσει τα δικαστήρια ότι είναι και συνταγματικό και συνάδει πλήρως με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είναι ένα κεφαλαίωδες εργαλείο για τον αγώνα κατά του εγκλήματος στο Ιλλανδικό νομικό σύστημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την ευκαιρία να λάβω το λόγο ενώπιόν σας και φυσικά είμαι έτοιμος να απαντήσω τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Κυρία Κόρκοραν. Υπενθυμίζω ότι έχουμε ακόμη ένα σημείο στην μέση διάταξη πριν τις 12.30, άρα 15 ε, λεπτά μένουν. Ε, κάποιος που θέλει να κάνει ερώτηση και εμένα, κυρία Ζήπελ, παρακαλώ δύο λεπτά. Προσπαθώ να είμαι σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Δεν με έπεισε αυτό που είπε ο κύριος Κόρκοραν. Αν υπάρχουν αποφάσεις ότι κάποιος έχει συσσωρεύσει ε, περιουσιακά στοιχεία λόγω εγκλήματος, το καταλαβαίνω. Αλλά από ό,τι κατάλαβα αυτά που είπε ο κύριος Κόρκοραν, δεν υπάρχει νομική απόφαση, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση. Εμένα μου φαίνεται ότι αναστρέφονται τα πράγματα, ότι γίνεται πρώτα η καταδίκη και μόνο μετά έχει κανείς το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενώπιον δικαστηρίου. Αυτό μου φαίνεται εντυπωσιακό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, υπάρχει μια αρχική υποψία και γίνονται αυτές οι διαδικασίες ή πηγαίνουν οι αρχές και κοιτάνε δεξιά τους λογαριασμούς να δουν αν υπάρχει κάτι το οποίο τους φαίνεται αξιοπερίεργο και μπορεί να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο μια απόφαση. Ποιος πρέπει να έχει την απόδειξη ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Όποιος έχει μια υποψία μπορεί πάντα να ξεκινήσει την ποινική διαδικασία και να δει κατά πόσον έχουν γίνει αυτές οι εγκληματικές ενέργειες. Όλα αυτά λοιπόν που λέει δεν μου φαίνεται να, δει, να συγκροτούν μια πολύ καλή διαδικασία. Μορβάη, δύο λεπτά. Σχετίζεται το ερώτημά μου με το προηγούμενο. Είπατε στην παρουσίαση ίσως ότι το ανώτατο το σταγματικό δικαστήριο έλεγξε, επαλήθευσε ε, σε σχέση με εγγυήσεις για ποινική διαδικασία για, αυτή, για αυτά τα, τους προσόδους αυτές και η απάντηση ήταν ότι δεν χρειάζεται και τα λοιπά, ότι μπορεί να είναι αστική η διαδικασία. Δεν ξέρω, μήπως δεν κατάλαβα πολύ καλά. Τι είπε το δικαστήριο πάντως. Μήπως και ο νόμος είναι υπό ε, εξέταση για αναθεώρηση. Το θέμα είναι το εξής. Το δικαστήριο έχει επιβάλει κάποια ελάχιστα πρότυπα για μια δίκαιη δίκαιη αντιμετώπιση. Είναι σαφές το ερώτημά μου. Κύριε Λάτφορ, δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ για την παρουσία την εκτίμηση ιδιαίτερω. Είναι πάνω το σύστημα και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά, φυσικά και εξαρτάται από το να εμπιστεύεται κανεί στα δικαστήριά του και αυτά θα εφαρμόσουν και τους νόμους. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό που θέλουμε να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα μπορούσε να είναι η δικαιολογία να αναλαμβάνεται δράση ε, μέσω του η δυνάμει του αστικού δικαίου. Και το θέμα είναι ή αφήνουμε κάποιους να ξεφεύγουν και να μπορούν να ζουν με περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτήσει από εγκληματικέ δραστηριότητε δεν μπορούμε να τα καταδικάσουμε ή είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα μέτρα που λαμβάνουμε εξασφαλίζοντας ε, όλα τα χέγγια τα οποία μας ε, περιγράψετε κι εσείς, για να μπορέσουμε να έρθουμε σε αυτές τις πρόκλησεις. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε πρώτα απ' όλα να έχουμε και να μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε όλα τα εθνικά νομικά συστήματα. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα ε, μαφιόσικου εγκλήματος και βέβαια των τεράστιων προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που μέχρι τώρα μένουν ατιμόρυτοι όλοι αυτοί που ζουν με αυτά τα χρήματα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο, το ε, Δικαστήριο του Στρασβούργου έχουν στην ομολογία τους εξηγήσει πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα, πιστεύω. Άρα θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στα μέτρα αυτά. Αυτό βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το τι μπορεί κανείς να εισάγει μέσω της οδηγίας που προτείνεται. Αυτό είναι ξεχωριστό θέμα δηλαδή για το εύρος, το νομικό εύρος των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, σε ό,τι αφορά την κατάσχεση των περισσότερων στοιχείων, αυτό το οποίο ισχύει στην Ιρλανδία απέδειξε ότι λειτουργεί ο σύστημα και μας έδωσε ε, και το δικαστήριο πολύ προσεκτικές ε, τιμιγορίες και αποφάσεις. Ο κύριος Βος, δύο λεπτά. Ο κύριος, ο κύριος Βος, δύο λεπτά. Έχω ένα θέμα βασικού χαρακτήρα σε σχέση με τη νομική βάση για τη διαδικασία. Στη Γερμανία έχουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ αστικών υποθέσεων και ποινικών υποθέσεων. Και γι' αυτό το ερώτημά μου. Καταρχήν, θεωρείτε ότι μπορεί ένα τέτοιο σύστημα όπως έχετε στην Ιλλανδία να εφαρμοστεί και σε διαφορετικά νομικά συστήματα χωρίς να υπάρξει κάποια προσαρμογή. Και δεύτερον, εγώ δεν καταλαβαίνω τη λογική που χρησιμοποιείτε ότι δεν μπορούμε να διώξουμε κάποιον ποινικά, δεν έχουμε καμία απόφαση από δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να κολλαστεί αυτός ο οποίος έχει κάνει αυτή την ε, ε, ενέργεια, την εγκληματική ενέργεια. Μα πού βρίσκεται η δικαιολογία που λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει το τεκμήριο αυτό, τόσο γιατί κάπου έχουμε ανθιστεί ότι κάποιος έχει πάρει τα λεφτά αυτά από κάποια εγκληματική ενέργεια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική σας σε αυτό το σημείο και δεν μπορώ να καταλάβω σε, μια, σε ένα νομικό πλαίσιο να δημιουργήσει νομική επιχειρηματολογία ώστε να ανατρέψει τελείως τη φυσική σειρά των πραγμάτων. Κύριε Κόρκορα, θέλετε να κάνετε μια σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε κι άλλο ένα σημείο στη μέση διάταξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω όσο το πιο σύντομα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, οι υποθέσεις που αναλαμβάνουμε ε, έχει προηγηθεί για αυτές ε, μεγάλη έρευνα. Δεν αναλαμβάνουμε ελαφρά ή βιαστικά τις υποθέσεις αυτές, χωρίς να έχουμε εξετάσει όλα τα στοιχεία προηγουμένως. Σε κάθε μεμονωμένη υπόθεση έχει προηγηθεί έρευνα, εκτεταμένη και διεξοδική. Πρέπει το δικαστήριο να πιστοποιήσει και να ε, βεβαιωθεί ότι μιλάμε για ε, προϊόντα εγκλήματος. Αυτό ε, πρέπει να το αποδείξει το δικαστήριο, να το δεχτεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστικό δίκαιο το οποίο χρησιμοποιείται αυτό, έχει να κάνει με το πρότυπο για το βάρος απόδειξης, για την απόδειξη. Πρόκειται για μια δράση in rem, κατά της περιουσίας και όχι κατά κάποιου ατόμου συγκεκριμένου, ούτε ε, επηρεάζει τα δικαιώματα κάποιου ανθρώπου. Είναι μια δράση in rem κατά, για, την περιουσία, για ένα περιουσιακό στοιχείο, εφόσον αποδειχθεί επαρκώς ότι άμεσα ή έμεσα αυτό το αγαθό αποτελεί προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος. Ε, πιο σύντομα δεν μπορούσατε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καταλάβαμε το νόημα. Αυτό αφορά βέβαια και τη δέσμευση και δίμευση πρώτων εγκλήματος, ε, που, ε, την έκθεση την οποία είχε αναλάβει η κυρία Μακοβέη. Και τις οργανικές διαπραγματεύσεις και σε ό,τι αφορά το Eurodac ε, έχει αναλάβει πάλι την έκθεση αυτή η κυρία Μακοβέη Πέντε λεπτά έχουν μείνει βέβαια. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να σας ε, δώσουμε και λίγα παραπάνω λεπτά για να μας κάνετε αυτή την παρουσίαση, κυρία Μακοβέη, πώς έχει κατάσταση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο δεύτερος τρίλογος για το Γιούντακα έγινε στις 7 Φεβρουαρίου. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παρουσίασαν τις θέσεις τους για τις ε, επίμαχες διατάξεις. η πολιτικά ε, επίμαχες διατάξεις ήταν η σήμανση των δεδομένων, άρθρο 18, οι υποθέσεις πρόσβασης στην Eurodac για λόγους επιβολής του νόμου, για, από τις αρχές επιβολής του νόμου, άρθρο 20, το ίδιο αντίστοιχο πρόβλημα στο άρθρο 21 για την πρόσβαση της Europol, δικαιώματα ενημέρωσης ε, του υποκείμενου των δεδομένων άρθρο 29, η αιτιολογική σκέψη 26 για την πρόσβαση και η αιτιολογική σκέψη για την πρόσβαση στις αρχές στις διοκτικές αρχές. Ό,τι αφορά την σήμανση, προτείναμε να επιτρέπεται σήμανση για σκοπούς ασύλου, αλλά να μην υπάρχει τέτοια πρόσβαση στις διοκτικές αρχές. Ζητήσαμε να υπάρχει ορισμός της σήμανσης, ε, τουλάχιστον σε αιτιολογική σκέψη, κατόπιν το Συμβούλιο εξετάζει ότι, ε, θεωρεί ότι η πρόσβαση στις αρχές επιβολής του νόμου είναι ουσιαστικού χαρακτήρα και δεν δέχθηκε τις ε, προτάσεις του Κοινοβουλίου. Μιλώ για τα άτομα που, λαμβάνουν, που έχουν λάβει διεθνή προστασία. Η Επιτροπή πρότεινε μια συμβιβαστική λύση να υπάρχει σήμανση μόνο για τις αρχές επιβολής του νόμου αλλά όχι για τη σήμανση αυτή καθεαυτή. Συνεχίζουμε να έχουμε τεχνικές συναντήσεις και συναντήσεις με τους κοιοδησίγητες. Πριν από λίγες έγινε τελευταία. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Έτσι όπως είναι η κατάσταση καλύτερα να μην πω πολλά. Ευχαριστώ. Σχόλια. Αν όχι, διακόπτουμε και θα συνεχίσουμε μετά το γεύμα στις 3. Μετά το